Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de commission des budgets. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας εδώ στην Επιτροπή των Προπολογισμών. Πρώτη συνεδρίαση μετά το καλοκαίρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους ξεκούραστους. Έχετε όλοι ένα ωραίο χρώμα, είστε μαυρισμένοι. Ελπίζω λοιπόν ότι καταφέρατε να ευχαριστηθείτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και ότι έχετε ξεκουραστεί και ότι έχετε πλέον ανακτήσει νέα δύναμη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα, τη ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που έχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών. Ονειρεύτηκα και κάτι κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτών ονειρεύτηκα ότι ήμασταν σε θέση να βρούμε τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να εξορροπήσουμε δαπάνες και έσοδα στον προπολογισμό. Προκειμένου να καταφέρουμε να εξαφανίσουμε στο τέλος κάθε οικονομικού έτους όλες αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες δεν έχουμε καταβάλει ως πληρωμές. Να καταφέρουμε λοιπόν να δώσουμε το κατάλληλο παράδειγμα ως Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την δημοσιονομική διαχείριση. Να καταφέρουμε δηλαδή να εξορροπούμε πάντα υποχρεώσεις, πληρωμές, έσοδα και δαπάνες. Ότι θα καταφέρνουμε επίσης ονειρεύτηκα να πετύχουμε μία συνένεση προκειμένου να βρισκόμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα, πιο κοντά στις πραγματικές δημοσιονομικές ανάγκες και πιο μακριά από ουτοπίες ή ψευδεστήσεις. Με όλα αυτά λοιπόν, ελπίζω ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να καταφέρουμε καταρχάς να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης, η οποία θα συνεχιστεί και το απόγευμα στις 3 το μεσημέρι. Όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς για τη σημερινή συνεδρίαση, είναι γνωστό. Το βλέπετε το γλωσσικό καθεστώς στο ενημερωτικό φυλάδιο του newsletter της Επιτροπής Προπολογισμών. Ελπίζω επίσης ότι έχετε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 7ης, 14ης και 23ης Ιουλίου και ελπίζω τα πρακτικά αυτά ανταποκρίνονται πιστά στα όσα είπαμε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών. Να προσθέσω επίσης κάτι. Πριν από λίγο ελήφθη μία απόφαση, κατά τη διάρκεια δηλαδή της συνεδρίας των συντονιστών, Και θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω και για αυτό το λόγο συγγνώμη για το ότι ξεκινήσαμε καθυστερημένα τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είχαμε εκτενείς ε, συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών. Μάλιστα δεν ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση αυτή. Θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα μετά το τέλος των εργασιών της Επιτροπής μας. Σήμερα λοιπόν το πρωί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών αναφερθήκαμε στην ε, ακρόαση του Επιτρόπου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό και για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην ακρόαση του υποψήφιου αυτού Επιτρόπου και εγκρίναμε τρεις γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν προς τον υποψήφιο αυτόν. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν, οι οποίες αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά τις προσδοκίες των εκπροσώπων των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Οι ερωτήσεις αυτές σας διαβιβάστηκαν, τις έχετε μπροστά σας μάλιστα αυτή τη στιγμή. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές τον κοινοτικό προπολογισμό. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στο ζήτημα της ερμηνείας που θα δώσει ο υποψήφιος επίτροπος για το πώς θα μπορέσει να αναθεωρήσει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο μέλλον. Ξέρετε ότι βρισκόμαστε αρκετά, με, κοντά μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί σύντομα και θα ρωτήσουμε τον υποψήφιο λοιπόν επίτροπο έμπρακτα πώς μπορεί να υλοποιήσει την προσδοκία αυτή. Και η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζετε ότι από το ένα έτος στο άλλο οι ίδιοι πόροι, οι οποίοι ουσιαστικά απαρτίζονται από τους ε, δασμούς, τους τελωνιακούς δασμούς, είναι πόροι οι οποίοι τροποποιούνται κάθε φορά με τις νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχουμε με τις τρίτες χώρες. Να λοιπόν, ποια απόφαση λήφθη πριν από λίγο να υποβληθούν τα τρία αυτά ερωτήματα προς τον νέο υποψήφιο επίτροπο και έχουμε μια γενικότερη συνένεση ανάμεσα στην ομάδα των συντονιστών για να υποβληθούν, να κατατεθούν επίσημα τα ερωτήματα αυτά. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα του προπολογισμού 2015 θα μπορέσουμε να διαιρέσουμε, αν θέλετε, τη συνεδρίαση μας σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα μπορεί να αφορά το τρίτο τμήμα του προπολογισμού και στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα υπόλοιπα τμήματα του προπολογισμού για το 2015. Όσον αφορά το τμήμα υπαριθμών 3, πρωτού δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας, θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω από τον γενικό μας εισαγητή, από την κυρία Γκαρθιά Ζαμπάλ, να μας παρουσιάσει το δικό της έγγραφο εργασίας όσον αφορά την τοποθέτηση του Συμβουλίου για το τμήμα 3 πάντα του προπολογισμού και να μας παρουσιάσει επίσης και τα αποτελέσματα της δεύτερης προαξιολόγησης, πρώτης αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν ε, υποβληθεί όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, τη δράση δηλαδή που πρέπει να αναλυφθεί. Κυρία Εισηγήτρια, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα αισθήματα αυτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει η Εισηγήτρια. Πέρασε ένας μισδιακοπών, οπότε τώρα ξαναγυρίζουμε ε, είμαστε υπατμόν όσον αφορά αυτή την διαδικασία του προπολογισμού, οπότε θα πρέπει τώρα να αναλύσουμε την πρόταση του Συμβουλίου και να προετοιμάσουμε τις τροπολογίες ε, για τις επιτροπές από πλευράς και των ε, πολιτικών ομάδων, τόσο ώστε να ξεκινήσουμε τις καθεαυτού ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας παρουσιάσω αυτό το έγγραφο εργασίας όπου και έτσι όλοι οι συνάδελφοι της Επιτροπές μας να έχουν ένα έγγραφο στα χέρια τους, να έχουν μια σύνοψη για το ε, πώς βλέπει το Συμβούλιο την πρόταση της Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο χωρίζεται σε δύο μέρη πρώτα-πρώτα, το πιο ε, ας το πούμε επεξηγηματικό κομμάτι ε, και το δεύτερο είναι πιο πολιτικού χαρακτήρα και επίσης υπάρχουν και τα σχόλια της εισηγήτριας, της ομιλούσης για να σας πω και βέβαια όλα αυτά είναι μια σύνοψη των δεδομένων που είχα στα χέρια μου και σας ε, επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για την δική μας πολιτική θέση σύμφωνα με σε όσα κατέληξαν οι ε, πολιτικές ομάδες και ο τρίλογος του Ιουλίου. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων είπαμε ότι θα πρέπει να να γίνουν οι επενδύσεις σε όλους τους τομείς που και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και ότι θέλουμε να προχωρήσουν ε, για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να μπορέσουμε ό,τι αποθεματικά υπάρχουν να τα απορροφήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε αυτούς τους τομείς, τα στρατηγικά αντίστοιχα προγράμματα. Ε, αυτά όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις, τώρα όσον αφορά τις πληρωμές. Πρέπει τις οφειλές μας να τις ε, εξοφλήσουμε. Να υπάρξει επομένως επαρκής χρηματοδότηση για αυτό το σκοπό για το 2015. Και αυτά είναι ε, τα βασικά μήνυματα τα οποία θέλει να στείλει στο Συμβούλιο το Κοινοβούλιο. Βέβαια, να δούμε το εξή. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του τι λέει και του τι διατυπώνει εγγράφο μετά και κυρίως ε, διατυπώνει σε νούμερα το Συμβούλιο. Γιατί ε, είπαμε ότι όντω θα πρέπει ναι, να έχουμε ανάπτυξη, να επενδύσουμε, να βοηθήσουμε την απασχόληση. Όταν όμως έρχεται η ώρα να δούμε τι νούμερα προτείνουν, βλέπουμε ότι εκεί που θα πρέπει να έχουν υπάρξει αυξήσει. έχουμε πρόταση περικοπών. Αυτά. Έχουμε επίσης ε, για τις επιτροπές, ε, προτάσεις επιτροπής 572 εκατομμύρια λιγότερα και όσον αφορά αυτά για τις υποχρεώσεις και ε, στις πληρωμές επίσης έχουμε πάρα πολύ σημαντικές περικοπές και βλέπουμε επομένως ότι κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτή την χιονοστιβάδα των χρεών που έχει σωρευτεί. Πάντως έχουμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Αν κοιτάξουμε αυτές τις δύο δηλώσεις για τις πληρωμές που προέκυψαν από το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα 13 χωρών οι οποίοι είπαν ότι στον βωμό της συνένεσης ε, συμφωνούν με την πρόταση αλλά προειδοποιούν ότι το πρόβλημα των πληρωμών είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρούν ότι τελικά δεν θα υπάρξουν αρκετά χρήματα για τις πληρωμές στο μέλλον. Γιατί έχουμε μια ομάδα επίσης από άλλες εννέα χώρες που λένε ότι ό,τι και να γίνει ποτέ δεν θα διατεθούν περισσότεροι πόροι και θα τηρηθούν οι σχετικές οροφές, ανώρια τέλο πάντων για τις δαπάνες. Και θέλουν επομένως έστω και τεχνητά να ε, μείνουν οι πληρωμές κάτω από αυτό το ανώριο παρά το ότι θα μείνουν κάποιες οφειλές οι οποίες θα είναι ανεξόφλητες. Αυτά για τις προτάσεις του Συμβουλίου για κάθε κατηγορία, τα έχετε όλα αυτά, έχετε όλα τα δεδομένα. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για την κατηγορία 1α. Είναι από τις πιο σημαντικές για μας. Και επίσης έτσι ε, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις ε, επενδύσεις, τις σχετικές και οι περισσότερες από τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο αφορούν ακριβώς την κατηγορία αυτή. Επίσης, με τις προτάσεις αυτές το Συμβούλιο όχι μόνο λέει όχι στις δικές μας προτάσεις, όχι μόνο αντιφάσκει προς ε, τα ίδια του τα ε, λόγια, αλλά έτσι παραβιάζουν την συμφωνία που είχαμε κάνει σε σχέση με τις επενδύσεις, σε σχέση με την υποστήριξη προώθηση των σχετικών προγραμμάτων. Είχαμε πει για το 2014 και τη χρήση του 2015 και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε σε αυτή την περίπτωση ε, για ένα από τα λίγα, μια από τις λίγες υποσχέσεις που αποσπάσαμε εμείς ως ε, Κοινοβούλιο σε σχέση με το χρηματοδοτικό πλαίσιο γιατί ακριβώς είπαμε ότι θα υπάρξουν επενδύσεις για το 14-15 το απαιτήσαμε εμείς και το αποσπάσαμε το συμφωνήσαμε αλλά να τώρα που το Συμβούλιο δεν σέβεται τα συμπεφωνημένα Οπότε, έχουμε τώρα και την κατηγορία υπαριθμών 3 σε κάποια προγράμματα ε, που είναι πάρα πολύ βασικά, που και εκεί προτείνουν ε, περικοπές. Η Ευρώπη για, ε, για τους πολίτες, ε, καταναλωτές, ισότητα, δικαιώματα σχετικά κλπ. Είναι δηλαδή κάποια προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε και εδώ θα ε, προσέχουμε και εδώ θα πρέπει να πούμε όχι σε αυτές τις περικοπές. Γιατί δεν νομίζω ότι βοηθούν αυτές οι μικρές περικοπές σε τίποτα σημαντικές οικονομίες για θεσμικά όργανα. Όμως θέτουν εν κινδύνο αυτά τα προγράμματα τα οποία τόσο ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο. Επίσης πάμε στην κατηγορία 4 τώρα και εκεί έχουμε κάποιες ε, περικοπές που επίσης είναι και απαράδεκτες και ακατανόητες. Μα τι γίνεται, είναι σαν να μην έχει επίγνωση το Συμβούλιο του ότι στον σημερινό κόσμο επιβάλλεται η χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων που καλύπτονται από αυτή την κατηγορία. Επιβάλλεται η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που αφορούν την ε, επίλυση κάποιων κρίσεων. Πρόκειται για σταθερότητα, πρόκειται για ειρήνη, πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια που καλύπτουν αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ακατανόητη η στάση του Συμβουλίου. Έχετε εδώ όλα τα στοιχεία για τις περικοπές. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τις ε, περιφερειακές ε, ε, κοινοτικές υπηρεσίες η θέση Κομισιών και του Συμβουλίου για αυτές τις αποκεντρωμένες όπως λέγονται επιχειρήσεις, υπηρεσίες. Εμείς έχουμε υιοθετήσει κάποια θέση και είπαμε ότι δεχόμαστε μια περικοπή αρχική 5% όπως πρότεινε η Κομισιόν. Όμως δεν δεχόμαστε το παραπάνω 5% το οποίο μετά προτείνανε. Εμείς θα συνεχίσουμε τη ρότα της αρχικής μας πρότασης. Αξιολογήσαμε τις προπασκευαστικές δράσεις, τα πιλωτικά προγράμματα σχετικά με τις πληρωμές. Τα έχει αυτά το εγγραφό εργασίας και για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι ανακατηγορία ε, τα παραθέσαμε εδώ τα στοιχεία και αναδεικνύουμε τις περιοχές, συγγνώμη, τους τομείς όπου έχουμε τις μεγαλύτερες περικοπές. Και τελικά θα πρέπει να προσέξουμε ότι είναι και θέμα εσωτερικό του Συμβουλίου, και θα γίνουν ε, κάποιες ε, ζυμώσεις, αλλά να δούμε το σύνολο, το σύνολο των περικοπών και το σύνολο των πληρωμών θα τα ε, ζυγίσουν, τελικά ξέρουν αυτοί πώς τελικά θα τα βρούνε ε, και έχουμε την πλειοψηφία των κρατών μελών οι οποίοι ελπίζουμε να προσχωρήσουν σε ε, μια τελική συμφωνία για τις περικοπές, για τις χώρες των συνοχής, για την κατηγορία 1α όλα αυτά θα πρέπει να τα εξασφαλίσουμε και τελικά το σύνολο του ποσού για τις πληρωμές να είναι επαρκές και κατόπιν να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων για να καλυφθούν οι ανάγκες για τις ε, πιστώσεις των πληρωμών. Είπαμε ότι για τους διορθωτικούς προπολογισμούς ε, υπήρχε σχετική συμφωνία για τη χρήση του 2015 και είπαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν εξυπηρετήσουμε τις οφειλές, τα χρέη μας, τις, ε, τα χρέη μας τα παλαιότερα και μετά θα δούμε τι θα πληρώσουμε το 2015 ε, δεν είναι τόσο δύσκολο να το σκεφτεί κανείς αυτό, να υπολογίσει τι χρειάζεται επιμείναμε σχετικά με αυτό και θα συνεχίσουμε ακριβώς την ίδια κατεύθυνση και θα πρέπει από σχέδια παντός όλα αυτά να τα σκεφτεί το Συμβούλιο και να εγκρίνει ταυτόχρονα τους διορθωτικούς προπολίγους 2, 3 και 4 και έτσι να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε τις οφειλές μας ή κάποιες τέλο πάντων αρκετές από τις οφειλές της παλαιότερες για να μπορέσουμε να μπούμε στο θέμα των πληρωμών ε, για το 2015. Τέλος Σεπτεμβρίου ελπίζουμε το Συμβούλιο μπορεί να μας παράσχει περισσότερα στοιχεία για το τι θα γίνει ε, σήμερα σε σχέση με τις οφειλές και να, δούμε από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρεσβεύει και έτσι να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα εκταμείευσης των πληρωμών για τις μελλοντικές χρήσεις. Τώρα, ένα σύντομο σχόλιο όσον αφορά τα πυροτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. 29 Αυγούστου λάβαμε την δεύτερη αξιολόγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 82 προτάσει. Λέει 81 η Κομισιόν, γιατί εδώ πέρα ενοποίησαν δύο. Και αυτέ λοιπόν 81 προτάσει τη Κομισιόν, ε, 9 ε, είναι μια χαρά, 20 είναι δυνατόν να υλοποιηθούν εν μέρη, 38 από αυτέ τι προτάσει ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες ή από προγράμματα τα οποία ήδη τρέχουν και έχουμε δέκα από αυτές τις ε, προτάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα όσα πρέπει να ισχύουν για τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις και θα πρέπει να γίνει σχετική αξιολόγηση. Εγώ ανέκαθεν θεώρησα ότι ισχύει το, η αξιολόγηση των επιτροπών μας είναι πάρα πολύ βασικό και έτσι μπορούμε να δούμε κατά πόσον τα πολιτικά προγράμματα μπορούν να προχωρήσουν. Αυτά όμως έχουν ε, συμβουλευτικό χαρακτήρα και αν και οι πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, κάποια τέτοια δράση μπορεί να προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, ε, δεν, το, δεν την έχει προτείνει τότε όμως θα κάτι η πρόταση των πολιτικών ομάδων. Και έχουμε επομένω μετά αυτού του δύο γύρου 69 προτάσει και ε, στον πρώτο γύρο 81 μετά το δεύτερο γύρο επαφών. Οπότε τώρα ε, θα πρέπει να τηρήσουμε τα όρια ανακατηγορία, αλλά μην ξεχνούμε ότι πάμε για όλα τα πιλωτικά στα 40 εκατομμύρια και για τις καινούριε καινούργιες 50 εκατομμύρια και το συνολικό όριο, η συνολική οροφή φτάνει τα 100 εκατομμύρια και όλα αυτά επομένως περιορίζουν το συνολικό πακέτο ε, το οποίο θα καλύψει πιλωτικά προγράμματα και προπροσκευαστικές δράσεις και επομένως το σύνολο όλων των προτάσεων φτάνει τα 208 εκατομμύρια εγώ τέλη του μηνός θα διατυπώσω μία πρόταση με προτεραιότητες των επιτροπών μας, των πολιτικών μας ομάδων. Θα προσπαθήσω να τηρήσω αυτά τα ανώρια, αυτές τις οροφές και ελπίζω ότι με την πρότασή μου θα μπορέσουμε να όσα ε, πρεσβεύουν οι πολιτικές ομάδες και οι καθέκας των βουλευτές. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια για την σαφέστατη αυτή παρουσίαση. η οποία όντως μας επιτρέπει να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Μετά τις πληροφορίες αυτές μπορούμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ. Ο κύριος Φερνάντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους. και είμαι βέβαιος ότι θα είναι δυνατόν να δώσουμε απόδειξη εργασίας μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις όπως η συνάδελφος έκανε καλή δουλειά και θα ήθελα να τονίσω εξαιρετική δουλειά έγινε έγινε εξαιρετική δουλειά μέχρι σήμερα το πρόβλημα όμως δεν είναι στη συνένεση στο κοινοβούλιο το πρόβλημα συνεχίζεται να είναι το πρόβλημα στο Συμβούλιο μιλάμε για το 2000, τον προϋπολογισμό 2015, βρισκόμαστε το, στο 2014, πολύ λίγο αντανακλά το δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο 2014-2020. Είναι ανάγκη λοιπόν να αντανακλάτε αυτό και πρέπει σύντομα να αναφερθεί στη συζήτηση αυτό, ώστε να υπάρξει συγκεκριμενοποίηση της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και το ίδιο το Συμβούλιο το έχει καθορίσει αυτό και έχει συμφωνήσει για αυτή τη στρατηγική και για τους στόχους αλλά το να καθοριστούν οι στόχοι και να μην έχουμε τα μέσα, τα κονδύλια να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι πρόβλημα και θεωρώ ότι σημαντικό θα ήταν όλοι οι πολίτες να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι πρόβλημα αξιοπιστίας αυτό. Το Συμβούλιο δεσμεύεται και μετά δεν επομίζεται τις ευθύνες να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις. Και όταν μιλάμε για πληρωμές κάνουμε λόγο για ήδη πληρωμές που έχουν γίνει, πρέπει να έχουν γίνει φοιτητέ για το έρασμος, για τα πανεπιστήμια. Κάνουμε λόγο για την έρευνα επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάνουμε λόγο για επενδύσεις για τη συνοχή, οικονομική συνοχή και κοινωνική συνοχή. Και είναι απαράδεκτο να μην πληρώνονται αυτά τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να πούμε και είναι μια γλώσσα που όλοι αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν. Και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κάποια κράτη απαιτούν κάποια πράγματα και άλλοι, άλλα κράτη έχουν δημοσιονομική πειθαρχία και τι γίνεται. Το ίδιο το Συμβούλιο δεν επομίζεται αυτή την υποχρέωση για αυτή την πειθαρχία. Και αρχίζει να υπάρχει αμφιβολία για την νομιμότητα που μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση όταν υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα και όταν έχουμε πληρωμές που δεν είναι ικανοποιητικές και δεν υλοποιούνται, δεν εκτελούνται και υπάρχει πρόβλημα. Και όσον αφορά τους λογαριασμούς του Συμβουλίου, είναι περικοπές αυτές που βλέπουμε, απερι, ε, απαράδεκτες περικοπές, όταν έχουμε και το, ε, που είναι πολύ σημαντικοί για την απασχόληση και την ανάπτυξη και για το κεφάλαιο επιπλέον όπου για τις περικοπές που γίνονται στην έρευνα επίσης ε, και ελπίζω για αυτόν τον λόγο ότι θα καταφέρουμε στο τέλος να επιβάλλουμε την κοινή λογική στο Συμβούλιο και τα 13 κράτη-μέλη τα οποία είπαν ουσιαστικά επί της ουσίας ότι δεν είναι ε, διαθέσιμα για τις πληρωμές αυτές, επιπρόσθετες πληρωμές, όταν όμως κάνουμε λόγο για αυτόν τον προϋπολισμό του 2015 και για την αύξηση που λέει ότι υφίσταται και ότι υπάρχει το Συμβούλιο, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο του 2015 είναι μια μείωση, συρρήκνωση στον πραγματικό προϋπολογισμό του 2014. Διότι αν εξετάσουμε και λάβουμε υπόψη τον προϋπολογισμό του 2014 και επιπλέον και τους διορθωτικούς ε, ε, προϋπολογισμούς, πράγμα που δείχνει ότι δεν υπήρξε πειθαρχία από πλευράς του Συμβουλίου σε σχέση με την ύπαρξη, την αναγκαιότητα διορθωτικών προϋπολογισμών, τότε καταλήγουμε στο ότι ο προϋπολογισμός που είχε υπόψη το Συμβούλιο για το 2015, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το 2015 με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς ε, συνεπάγεται μια μείωση ουσιαστική για τον προϋπολογισμό του 2015 και πέρα από αυτό είναι σημαντικό να αντανακλάται αυτή η κατάσταση, η σημερινή κατάσταση, στην κατηγορία 4, αλλά και σε άλλες κατηγορίες επίσης, όχι μόνο για τη διεθνή ε, βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια που πρέπει να εκτελέσουμε, αλλά επίσης και την κατάσταση και το πρόβλημα που υφίσταται και είναι μια κατάσταση που ξύνεται στην Ουκρανία για παράδειγμα και για οποιασδήποτε εξηγήσει όσον αφορά για τον προϋπολογισμό του 2015 σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες όπως για παράδειγμα την κατηγορία 2 όπου έχουμε την Γεωργία συγκεκριμένα. Για όλους αυτούς τους λόγους από πλευράς μας θα συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο στην εισηγήτρια και θα την υποστηρίξουμε και θα την βοηθήσουμε ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια των πολιτών ε, δεσμεύσεις με τη στρατηγική του 2020 που πρέπει να επιτευχθούν και όπου στόχος μας είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η απασχόληση να μπορέσουν ε, πραγματικά να επιτευχθούν και να εκτελεστούν αυτές οι υποχρεώσεις. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Μάνκα. Σας ευχαριστώ. Πρόβλημα με το μικρόφωνο. Μικροφωνίζει. Δεν ακούγεται, μικροφωνίζει. Το βασικό πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε έχει να κάνει με τις πληρωμές. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία πέντε χρόνια πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές δυσκολίες καταβολής πληρωμών για πολλούς λόγους. Ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι ότι δεν καταφέρνουν οι επιχειρήσεις αυτές να λάβουν τα απαραίτητα δάνεια από τις τράπεζες ή από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Εγκρίναμε μια οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας ότι θα πρέπει οι ε, επιχειρήσεις να λαμβάνουν από το δημόσιο τα χρήματα τα οποία το δημόσιο τους οφείλει μέσα σε 30 μέρες το αργότερο. Βλέπουμε όμως ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να λάβουν τα χρήματα αυτά στο απαραίτητο χρονικό διάστημα. Επομένως θεωρώ ότι το 2015 και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Δεν θα έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψουμε τις ε, υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Εγώ όταν ήμουν δήμαρχος είχα αντιμετωπίσει ένα ανάλογο πρόβλημα. Για πάρα πολλούς μήνες δεν καταφθάνανε τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία χρειαζόμουν απαραίτητο προκειμένου να καταφέρω να υλοποιήσω κάποια προγράμματα τα οποία ήδη είχαν εγκριθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την υλοποίηση πάρα πολλών κοινοτικών προγραμμάτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται υπό έντονη πίεση αυτή τη στιγμή. Αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μη άλλο, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο συγκεκριμένη. Όταν φαίνεται ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ασφάλουν κατά τη χρησιμοποίηση των κοινωτικών κονδυλίων, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ακόμα πιο αυστηρή. Τα λέω όλα αυτά διότι συνειδητοποιώ ότι η μόνη λύση που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή είναι να καταλήξουμε σε μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των παραδοσιακών ιδιών πόρων. Αν δεν καταφέρουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό, κάθε χρόνο θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μεταρρυθμίσουμε αποτελεσματικά το σύστημα των ιδιών πόρων. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε θέσει ένα σχετικό ερώτημα στον υποψήφιο επίτροπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Στάντερ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Ε, για την Επιτροπή Δικαιωμάτων Καταναλωτών ε, είμαι εισηγήτρια όσον αφορά τον προϋπολογισμό και οπότε ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα των πυροτικών προγραμμάτων και θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που εξηγήσατε όλη αυτή τη διαδικασία για το πώς αυτά τα προγράμματα τα οποία προτείνει κάθε επιτροπή πρόκειται να διεκπαιριωθούν και να πάρουν το δρόμο τους. Επίσης μου ζήτησε η Επιτροπή μου ε, να σας εξηγήσω τι προτείναμε, τι έγινε τα ΜΜΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει όλα αυτά τα, ε, ε, να σας πω ότι οι πολιτικές ομάδες τα υπεστήριξαν στην Επιτροπή μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να δούμε πώς αυτά θα προχωρήσουν με έναν τρόπο ε, διάφανο και θα πρέπει η Επιτροπή μας να ε, παρακολουθεί εξελίξεις, να ασχοληθούν όσοι θέλουν με αυτά και το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε το πώς θα εξασφαλίσουμε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα ε, δημοσιοποιούνται και να είναι γνωστό επίσης ποια θα είναι η τύχη του κάθε υπηρετικού προγράμματος. Βεβαίω η Επιτροπή Καταναλωτών ε, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τις ε, εξελίξεις της σημερινής. Ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε τώρα το λόγο. Λέει ο πρόεδρος έχει ο κύριος Κόλμαν. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και από τη δική μας ομάδα ευχαριστούμε τη Γενική Συγήτρια πολύ για τις διεξοδικές παρατηρήσεις της. Πιστεύω ότι και επανειλημμένα αναφέρθηκε αυτό, ότι εμείς πράγματι έχουμε δύο διαφορετικές πτυχές που ε, ασχολούμαστε με αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού 2015. Αφενός έχουμε τις αδρές γενικές γραμμές, ε, τον όγκο ιδιαίτερα αυτού του προϋπολογισμού και αφετέρου για τα περιεχόμενα, για την ουσία. Αν δούμε τον όγκο καταρχήν του προϋπολογισμού πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα απλά και μόνο, ότι αυτοί οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο όγκος των πληρωμών αυξάνεται κατά κάτι παραπάνω από 1%. Αλλά αυτό ισχύει μόνο αν τα συγκρίνουμε αυτά τα ποσά με τον προϋπολογισμό του 2014 ακόμα και των συμπληρωματικών προϋπολογισμών που πρέπει να εγκριθούν. Δηλαδή αν πάρουμε τον προϋπολογισμό αυτό και τον συγκρίνουμε του 2014 με το 2015, τότε αυξάνεται το σύνολο κατά 5% αν πάρουμε τον αρχικό προϋπολογισμό του 2014. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού πιθανότατα έχουμε νέα αποθεματικά. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα σχέδιο που, όπως το λέμε, είναι ε, επί ε, ξηρού ακμής ας το πω έτσι και πρέπει εδώ να λάβουμε πάλι υπόψη το πρόβλημα το οποίο συχνά αντιμετωπίζουμε δηλαδή όσον αφορά τα ραλ, τα γέστα λικίντε, τα υπόλοιπα προσπληρωμές, προσπληρωμή. Αυτά τα υπόλοιπα προσπληρωμή προς εξόφληση αυξήθηκαν σημαντικά. Το 2000 ε, είχαμε 66 δις ευρώ. Το 2007 139 δις ευρώ και τέλος του 2013 222 δις ευρώ υπόλοιπα προς εκτέλεση. Το 2010 στο 2013 κατά 70 δις αυξήθηκαν αυτά τα υπόλοιπα προς πληρωμή. Και εκεί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να γνωρίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή την εξέλιξη πρέπει να την καλύψουμε και από πλευράς προϋπολογισμού. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Μαθηματικά υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε λοιπόν αφενός θα αυξήσουμε τους, τις πληρωμές στον προϋπολογισμό αυτών ή θα μειώσουμε μελλοντικά τις πιθανές υποχρεώσεις προς πληρωμή. Αυτή την αλήθεια, αυτό το συμπέρασμα που αληθεύει δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε Όλα τα άλλα δεν οδηγούν σε καμιά λύση. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι υπό αυτό το πρίσμα, υπό αυτή την πτυχή, τον προπολογισμό στι αδρέ γραμμέ, στι γενικέ γραμμέ πρέπει να τον επανεξετάσουμε και πρέπει να αποφασίσουμε προ μία κατεύθυνση. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε διαφορετικέ απόψει. Εμεί από πλευρά τη ομάδα μα, όταν λέμε ότι πρέπει να ε, υπάρχει μια πολιτική λιτότητα, τότε είμαστε κατά τη αύξηση ε, των πληρωμών ε, τότε αυτό τι θα σήμαινε για να είμαστε συνεπείς. Ε, ότι οι υποχρεώσεις θα πρέπει να μειωθούν, ώστε να υπάρξει μια αντιστάθμιση στα δημοσιονομικά από πλευράς προπολογισμού στο μέλλον. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε να επανέλθουμε στη δημοσιονομική πειθαρχία που πρέπει να αποκατασταθεί. Φυσικά υπάρχουν και επί της ουσίας κάποια θέματα που πρέπει να τα εξετάσουμε. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν ήδη. Για παράδειγμα, το θέμα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και οργανισμών, των οργανισμών και υπηρεσιών γενικά. Είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες και οργανισμοί αναγκαίοι και αναγκαίες. Πρέπει να το θέσουμε αυτό το ερώτημα όταν έχουμε υπηρεσίες και οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Να ρωτήσουμε γιατί τις χρειαζόμαστε ή τους χρειαζόμαστε. Ποια πρόσθετη αξία απορρέει από την ύπαρξή τους. Δεν μπορεί να αναμένει κανείς μια αύξηση αποτελεσματικότητας ε, στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν κάποια από αυτές οι υπηρεσίες οι οργανισμούς ε, καταργηθούν. Το ίδιο πιστεύουμε και για το προσωπικό, ότι πρέπει εκεί να υπάρξουν εξοικονομήσεις, όχι μέσω περικοπών μισθών του υφιστάμενου πληρωμού, ε, του υφιστάμενου ε, προσωπικού, αλλά όσον αφορά την μείωση των δαπανών, όσον αφορά το συνολικό αριθμό των στελεχών. Και σε σχέση με τον προϋπολισμό εκπλήσωμε κάπως ως νεοεκλεγής Ευρωβουλευτής. Στους λίγους μήνες όπου βρίσκομαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο προσπαθώ να ε, καταφέρω να αποκτήσω μια επισκόπηση. Τι γίνεται με αυτά τα 222 δις ε, ραλ υποχρεώσεων, rest λικιντέ υπολείπων προς εκτέλεση. Σε πόσα χρόνια θα μπορέσουν να καλυφθούν. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον προγραμματισμό των εργασιών μας αυτό και δεν είναι δεδομένο τώρα αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Με μεγαλύτερη διαφάνεια μπορούμε καλύτερα να πορευθούμε προς το μέλλον και να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Πρέπει να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία και να διατεθούν λοιπόν, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και μια τελευταία παρατήρηση. Σε όλες τις δαπάνες πρέπει, πιστεύουμε, πάντα να μπορούμε να εξετάσουμε αν η βασική σκέψη για την αρχή της επικουρικότητας μπορεί να λειτουργήσει που πάντα από όλα τα κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία παρουσιάζεται το σημαντικό επιχείρημα. Η επικουρικότητα λοιπόν διασφαλίζεται και εδώ υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δεν είναι απόλυτα αναγκαία υπό το πρίσμα των εθνικών κρατών αν θα μπορούσαν για παράδειγμα να χρηματοδοτηθούν από πλευρά τους. Πρέπει να δούμε, έχουμε τη σωστή κατεύθυνση εδώ, έχουμε το σωστό προσανατολισμό και νομίζω είναι δίκαιο και νομίζω νομιμοποιημένο να υπάρξει η διασφάλιση των επενδύσεων από πλευράς μας. Αλλά ερώτημα, τι είναι επενδύσεις. Υπάρχει εδώ ένα θέμα ερμηνείας, αν ε, κάποιες δαπάνες είναι σκόπιμες ή όχι και σε τι σκοπεύουν. Στη Γερμανία έχουμε κάποια παραδείγματα, για παράδειγμα το αεροδρόμιο στο Βερολίνο Πράγματι, αδημορώ να δω, θα μπορούν κάποτε να απογειωθούν αεροπλάνα από αυτό το αεροδρόμιο που τόσο καθυστερεί στο Βερολίνο. Με εξέταση των πραγμάτων θα υπάρξει πρόσθετη αξία υπέρ των πολιτών από τέτοιες δράσεις. Ευχαριστώ. Merci, Ο κύριος Τωρεβάτς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κι εγώ σχολιάζοντας τα όσα είπε η συγγήτρια η γενική περιγραφή των πραγμάτων που έκανε είναι μια περιγραφή με την οποία νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε περισσότεροι στην Επιτροπή μας και γενικότερα στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι ε, το Συμβούλιο έχει μειώσει πολύ περισσότερο τις πληρωμές από ότι τις υποχρεώσεις. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό τον οποίο προτείνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να αναλάβουμε εμεί τις ευθύνες μας και θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά τα πράγματα και από την πολιτική τους διάσταση. Εμείς οι πολιτικοί πολύ συχνά υποσχόμεθα πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε στην πράξη να κάνουμε και στη συνέχεια κατηγορούμε άλλους ανθρώπους για τη μη τήρηση των υποσχέσεων. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη φορά όσον αφορά τις, την ανάληψη υποχρεώσεων. Έχουμε από την άλλη και τη στάση του ίδιου του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο πολλές φορές ακολουθεί απλώς μόνο την πολιτική των κυβερνήσεων χωρίς να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μειώνε λοιπόν τις πληρωμές και πολύ συχνά, χωρίς να γνωρίζουν πολύ καλά κάποιε βασικέ έννοιε των μαθηματικών δημιουργούν μια μη βιώσιμη κατάσταση. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θέλει να αυξήσει τι πληρωμέ για κάποιε γραμμέ του προπολογισμού που θεωρείται είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Παράλληλα όμω θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που δίνουμε νέε υποσχέσει, που αναλαμβάνουμε νέε υποχρεώσει. Δεν μπορούν αυτέ πλέον στο μέλλον να είναι ιδιαίτερα υπερβολικέ ή να μην είναι ρεαλιστικέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν πραγματικό προπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο να μην έχει πλέον ανεξόφλητε αιτήσει πληρωμών όπως ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τα κράτη-μέλη, όπως είπε και ο συνάδελφος Φερνάντες. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές σε αγαπημένα σημεία που έχουμε στον προπολογισμό. Το Συμβούλιο, από την άλλη, θα πρέπει βέβαια να σταματήσει να εμένει τόσο πολύ στη θέση του. Οι περικοπέ επηρεάζουν το 1, 4, το 1α και το 4, οι περικοπές του Συμβουλίου. γραμμέ του προπολογισμού που είναι πολύ σημαντικέ για μας, τμήματα του προπολογισμού που αποτελούν προτεραιότητες. Στο 1α θα είχαμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την πρωτοβουλία για τους νέους και να οδηγήσουμε σε νέες θέσεις εργασίας, καθώς επίσης σε απασχόληση, σε καινοτομία και ανάπτυξη. Αν δεν καταφέρουμε να προωθήσουμε την πρωτοβουλία αυτή για την απασχόληση, δεν θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε και τις επιχειρήσεις προκειμένου να είναι καινοτόμες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και νέες ευκαιρίες για τους νέους. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας κουράσω με όλη την ανάλυση της ε, αλυσίδας αξίας αν θέλετε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τη βιομηχανική διάσταση των πραγμάτων. Όσον αφορά το τμήμα 4, έχουμε την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη... έχουμε επίσης τη χρηματοδότηση προς τις χώρες της Αφρικής καθώς επίσης και προς την Ουκρανία. Ήμουν ανταποκριτή στη Ρωσία στο παρελθόν και γνωρίζω πραγματικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πραγματικά ακολουθεί μια εντελώς λαθασμένη πολιτική. Έχουμε όμως και στην Ουκρανία πολύ σημαντικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή η ε, Ουκρανία ζητά από εμά μια υποστήριξη που θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε εμεί να παρέχουμε. Όχι μόνο προ τι συμβουλέ που μπορούμε να δώσουμε, αλλά και προ τη χρηματοδότηση που μπορούμε να παρέχουμε προ την Ουκρανία. Επίση, έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη στον προπολογισμό 2014 όσον αφορά τον προπολογισμό 2015. Ελπίζω ότι θα καταφέρει το Συμβούλιο να εγκρίνει τον τελικό αυτό προπολογισμό χωρί να έχουμε δραματικέ καταστάσει όπω η τελευταία πράξη στην Τόσκα, για παράδειγμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλου στρατινισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Ο παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σαφές έγγραφο εργασίας, όπου πολύ καλά επεξηγούνται πού βρίσκονται τα προβλήματα. Και σαφώς γίνεται αναφορά στην μη συνεπή θέση του Συμβουλίου είναι σημαντικό αυτό σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ε, που εκκρεμούν. Η κατεύθυνση που ακολουθείται από το έγγραφο εργασίας είναι εξαιρετική πιστεύω. Και για ένα νέο Ευρωβουλευτή που εκπλήσεται για την μη συνέπεια, για τις ασυνεπείς ε, θέσεις που πολλές φορές υιοθετούνται, αυτό που διαρωτώ με είναι αν όλα αυτά τα δούμε και αν μπορούν να επαναληφθούν όλα αυτά και του χρόνου για άλλη μια φορά. Προσπαθώ να διαρρήξω αυτό το φαύλο κύκλο ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια πρόοδος που θα μπορέσει να επιτευχθεί. Διότι στις διαβουλεύσεις, στις διαπραγματεύσεις πρέπει να ακολουθήσουμε το στόχο να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Και το Συμβούλιο θα πρέπει για παράδειγμα από πλευράς του τα πολιτικά δημοσιονομικά θέματα να τα λάβει υπόψη. Είναι μια καλή σύσταση αυτή για το Συμβούλιο. Οι κατηγορίες δεν δίνουν πάντα ε, τη διαφάνεια που απαιτείται. Υπάρχουν ε, θέματα που είναι απόλυτης προτεραιότητας, ανεργία νέων, προγράμματα για την έρευνα για παράδειγμα, που πρέπει να τύχουν προτεραιότητας. Η έρευνα οικονομικά και κοινωνικά. Είναι σημαντική η έρευνα. Η έρευνα είναι σημαντική και για το μέλλον των παιδιών μας. Αλλά αυτό που για τις επενδύσεις προσέχουμε επανειλημμένα είναι ότι εθνικά σχέδια και ευρωπαϊκά σχέδια δεν ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ τους. Πρέπει να δει κανεί ε, ποιες τάσεις είναι διασυνοριακές και ως Κοινοβούλιο πρέπει να σκεφτούμε πού θα θέσουμε προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Η κυρία Νιρέντα έχει το λόγο. Και εγώ να συμφωνήσω με την εισηγήτρια. Συμφωνώ στα όσα είπε για τα πυροτικά προγράμματα όλοι εδώ. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να τιμούμε τις δεσμές μα και τις πιστώσεις άρα υποχρεώσεων και θα πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτο το να μην εξυπηρετηθεί ε, η υπόθεση των οφειλών μας και άρα θα πρέπει να προσέξουμε τις επενδύσεις και δεν θα πρέπει ε, για τις πιστώσεις υποχρεώσεων να έχουμε και άλλες ε, περικοπές. Θα πρέπει οι δεσμεύσεις μας να τιμηθούν, να καλυφθούν. Να οι υποσχέσεις μας και ε, είπαμε ότι θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και όχι άλλες ε, περικοπές. Αυτό και ιδίω εμάς στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όσον αφορά για ε, την περικοπή του προσωπικού σε σχέση με τόσα είπε κάποιος. Εγώ μιλώ κελτικά, ιρλανδικά, έχει αναγνωριστεί η γλώσσα μας ε, ως γλώσσα εργασίας επίσημη. Δεν έχουμε όμως ούτε καν στην Ολομέλεια διερμηνία από την γλώσσα μας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν χωρεί μείωση, μάλλον αύξηση. Merci, madame. Monsieur... Ο Πρόεδρος, θα σε ευχαριστώ. Κύριος Βόν. This committee talks a lot about commitments and obviously commitments. Μιλούμε για αυτέ τι πιστώσει υποχρεώσεων που φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικέ οι υποχρεώσει μα, οι δεσμεύσει μα και βέβαια και οι πληρωμέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ για το Συμβούλιο και αυτό έχει ε, ε, καταδειχθεί τα τελευταία χρόνια που δεν θέλει, δεν θέλει το Συμβούλιο να καταβάλει αυτά τα οποία χρειάζονται για τι ε, πιστώσει υποχρεώσεων. 3,3% μας λέει ότι έχει γίνει αύξηση έτσι μας λέει και άρα θα λένε ότι θέλουν να δώσουν τόσο πολλά. ή όχι, εμείς όμως ε, έχουμε άλλη βάση υπολογισμού και άρα καταλήγουμε σε άλλα νούμερα για τους προϋπολογισμούς και ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα για τις πληρωμές και ξέρουμε ότι τέλος της παρελθούσης χρονιάς μας είπε η Κομισιόν ότι είχαμε ε, να, να, να εκκρεμούν 23 ε, δις ευρώ. Οπότε και εμείς τα υποδείξαμε αυτά τα προβλήματα, δεν δώσαν σημασία για όλα, όλα αυτά τα, τα, τα χαρέ, αυτές τις οφειλές οι οποίες ακόμη κρεμούν. Και είδαμε τι γίνεται με, ε, με κάποια προγράμματα, με πανεπιστήμια, με επιχειρήσεις λοιπόν, με οργανισμούς, φορείες οι οποίοι έχουν πληγεί πάρα πολύ, διότι καθυστερούν πάρα πολύ οι δέουσες πληρωμές να εκταμιευθούν. Οπότε ε, θα πρέπει να μας ακούσουν. Εμείς τα προβλήματα αυτά τα επισημαίνουμε ε, υπάρχει έλλειψη στενότητας κλπ. Αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους φορείς, επιχειρήσεις και κλπ. Άρα θα πρέπει να δούμε με συγκεκριμένα ε, στοιχεία τι γίνεται με την κάθε των εκταμιεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Γενική Εισηγήτρια που μας παρουσίασε εξειδικευμένα την κατάσταση ως έχει για τον προϋπολογισμό. Έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που δεν έχει σαφή, σαφή στόχους και μια στρα, σαφή στρατηγική για κάθε μια από τις κατηγορίες δημοσιονομικά. Δεν αναγνωρίζουμε λοιπόν σαφώς τους στόχους της, ε, των δημοσιονομικών γραμμών αυτών, των κονδυλίων αυτών. Επιπλέον δεκάδες πληροφορίες έχουμε, αλλά πέρα από αυτά τα δημοσιεύματα από πλευρά ε, τύπου, δεν γνωρίζουμε αν τα κονδύλια τα οποία έχουν επιμεριστεί είναι επαρκή ή όχι ή και σε ποιο μέτρο θα μπορέσουν ε, να δαπανηθούν και αυτές οι πληρωμές θα είναι καθοριστικές θα ε, ψηφίσουμε ένα προπολογισμό του 2015 χωρίς να γνωρίζουμε τους άλλους επιτρόπους και ποιε είναι οι ιδέες τους και η στρατηγική τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιτροπή χωρίς να υπάρχει πολιτική υποστήριξη και αρρωγή επιβαρύνονται εδώ γραφειοκρατικά τα πράγματα από το Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καμιά πραγματική επαφή με την πραγματική ζωή μεταξύ αυτών των σχεδίων. Δαπανώνται εκατομμύρια χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει με τους στόχους. Για τα πιλωτικά προγράμματα θα ήθελα να πω δύο λόγια για την αξιολόγηση ενός προγράμματος για την υγειονομική κατάσταση και περίθαψη του, του κόσμου της υπαίθρου. Σημαντικό αυτό ε, για μας. Και υπάρχει και ακόμα ένα άλλο πολι, ε, πιλωτικό σχέδιο που δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα. Για όλα αυτά τα σχέδια τα οποία είναι συναφή, τα αποτελέσματα και οι αξιολογήσεις είναι διαφορετικές και διαφορετικά. Πώς γίνονται λοιπόν αυτές οι αξιολογήσεις διαρωτώμεθα για τέτοιου είδους προγράμματα. Πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος σαφών κριτηρίων για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα οπωσδήποτε και εκ προημίου θα πρέπει να πούμε ή θα πρέπει να δεχθούμε το α ή το β και στη συνέχεια τα υπόλοιπα τα συνεπαγόμενα ή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από πλευράς πλειοψηφίας ευρωβουλευτών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και έτσι θα έχουν δικαίωμα να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Ολμάιερ έχει το λόγο. Η κυρία Χολμάιερ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν κάποιες παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Θα μπορούσα να πω και ίδια, η ίδια διαδικασία όπως την γνωρίζουμε κάθε χρόνο ακολουθείται εδώ και πέντε χρόνια τώρα περίπου. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις από ό,τι πληρωμές. Και αυτό το πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια είναι πρόβλημα. Και αυτό παραμένει και διαιωνίζεται ως πρόβλημα και δεν τροποποιείται, δεν αντιμετωπίζεται με κάποια συνέπεια. Και δυστυχώς έχουμε και την ίδια δομή, το ίδιο πρόβλημα και στα πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα. Και αυτό το πρόβλημα επιβαρύνει και θα ήθελα να πω ότι αμφιβάλλω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί αποτελεσματικά. Εδώ λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον προϋπολογισμό κινούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Ένας τέτοιος προϋπολογισμός όταν έτσι καταρτίζεται πρέπει να μας κάνει να διαρωτηθούμε και να θέσουμε ερωτήματα. Δεν είναι ο συνηθισμένος, ο συνήθις τρόπος να, να καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός έτσι. Αν θέλουμε να λειτουργεί ένας προϋπολογισμός όπως το θέλουμε και να μπορούν να καταβληθούν κονδύλια και ποσά όπως πρέπει, ε, τότε δεν πρέπει να ακολουθείτε μια τέτοια διαδικασία. Μετά επίσης αυξάνονται διαρκώς τα υπόλοιπα και όταν έχουμε 24 δις τώρα στα οποία έχουμε καταλήξει, το μέγεθος των πληρωμών από τους τελευταίους προϋπολογισμούς ή των, ε, ε, των εξοφλητικών από τους προηγούμενους προϋπολογισμούς περιορίζουν διαρκώς το περιθώριο και διαρκώς μας πιέζει αυτή η κατάσταση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επανειλημμένα αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη νομική βάση. Η νομική βάση που έχουμε μπορεί ένα τέτοιο θέμα στο Συμβούλιο να αφήνει ελευθερία απόφασης και ε, κατά διακρι... στη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει το Συμβούλιο. Πώς είναι δυνατόν ε, να υπάρχει η έγκριση ε, πληρωμών και μετά η μη καταβολή πληρωμών. Πρέπει να δούμε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει το δικαίωμα να αναβάλλονται οι εξοφλήσεις πληρωμών και η καταβολή κονδυλίων που πρέπει να καταβληθούν. Έχει δίκιο ο συνάδελφος που λέει ότι όταν οι κοινότητες υποχρεούνται μέσα σε 30 ημέρες να εξοφλούν λογαριασμούς και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει εξαίρεση, είναι ενδιαφέρον να ρωτήσουμε και να δούμε γιατί το Συμβούλιο ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση και διαφορετική πορεία και δεν εξοφλεί λογαριασμούς μέσα σε 30 ημέρες ή έστω και μέσα σε μια μεγαλύτερη προθεσμία όπως σε σχέση με εταιρείε για παράδειγμα. Είναι προβληματική αυτή η κατάσταση το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα διότι όλο και περισσότερο αυτή η κατάσταση θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Αυτό είναι μια εκ παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Και επιπλέον από πλευράς του, τον, του κέντρου βάρους όταν περικόπτονται κονδύλια από την έρευνα πρέπει να προβληματιστούμε. Δεν πρέπει να επιλέγεται πάντα η έρευνα και εκεί να περικόπτονται τα κονδύλια γιατί χωρίς ε, την έρευνα δεν θα υπάρξει μέλλον για την Ευρώπη, όπως και σε άλλους τομείς. Και υπάρχει, θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ανταγωνιστικότητα για μας και όχι να αφαιρούμε την ανταγωνιστικότητα αυτήν περικόπτοντας την έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφαιρούνται θέσεις απασχόλησης από την Ευρώπη, να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα και να καταλήγουμε σε προβλήματα οικονομικά και δημοσιονομικά ως Ευρώπη. Κάποιες παρατηρήσεις επιτρέψτε μου να κάνω για τον προϋπολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρότι σε σχέση με το βάρος, ότι το βάρος αυτού του προϋπολογισμού δεν είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με άλλους προϋπολογισμούς, παρόλα αυτά κάποιες παρατηρήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου τις επόμενες δύο εβδομάδες διακόπτει ο Πρόεδρος. Κυρία Χολμάιερ, θα επιστρέψουμε στο σημείο αυτό όταν συζητήσουμε τα υπόλοιπα τμήματα του προπολογισμού. Α ολοκληρώσουμε πρώτα τη συζήτηση για το τμήμα 3. Εντάξει, μία μόνο παρατήρηση για τα πιλωτικά προγράμματα. Στα πιλωτικά προγράμματα πρέπει ειλικρινά να πω ότι μόνο με την κατηγορία Α ε, επαρκούμεθα η κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αμφισβητήσιμη και δημιουργεί ερωτήματα. Είμαι ειλικρινής και μιλάω ανοιχτά. Τώρα, για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα μπορούσε να βοηθήσει ε, και δίνει μια αξιολόγηση α όταν υπάρχει συμμετοχή των Ευρωβουλευτών, αν δεν υπάρχει αυτή τότε παίρνει Β ή Γ, B ή C ως ε, βαθμό. Θα πρέπει ως βουλευτές να δούμε πώς θα θέσουμε προτεραιότητες για αυτό το πεδίο και μετά να σκεφτούμε πώς θα έχουμε προτάσεις που θα αντιμετωπιστούν ε, με τον ε, εύθετο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εδώ έχουμε συναδέφους άλλων επιτροπών που έχουν εξαιρετικές ιδέες για πιλωτικά προγράμματα και υπάρχουν εδώ αποτυχίες επειδή δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα επαναλαμβάνεται για πέμπτη φορά για παράδειγμα το εγχείρημα και ε, ε, είχαμε κάτι το οποίο υποστηριζόταν από το όνομα ενός Ευρωβουλευτή. Θα ήθελα να είμαστε πιο ευσυνείδητοι με τέτοιου είδους πιλωτικά προγράμματα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντελάνο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία την οποία έχει κάνει. Νομίζω ότι ε, πολλά σημεία σωστά υπόθηκαν από αυτήν. Θα ήθελα όμως να πω ότι ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριφερόμαστε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στα τέλη Μαΐου του 2014. Εξελέγει ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύντομα θα έχουμε και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεπώς θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα νέο προσανατολισμό όσον αφορά την Ευρώπη. Ένας νέος προσανατολισμός που ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει να δώσουμε πλέον ένα τέλος στην κρίση και στη λιτότητα. Η προεκλογική εκστρατεία μας επέτρεψε να έρθουμε πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι μας είπαν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να λαμβάνει δράση κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Συνεπώς εμείς, όντας το μόνο θεσμικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, οφείλουμε πραγματικά να εκπροσωπούμε τη φωνή αυτών των πολιτών, <laughs> κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ήμουν επικεφαλής περιφέρειας στο παρελθόν στη χώρα μου και συντοπιώ ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο τα ταμεία αυτά καθώς επίσης και το ρόλο μόχλευσης που έχουν. Αν δεσμευόμαστε λοιπόν να χρηματοδοτούμε κάποια έργα, κάποια προγράμματα και στη συνέχεια δεν μας σε θέση να εξοφλήσουμε τις τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις δηλαδή που έχουμε αναλάβει, τότε υπάρχει πραγματικό πρόβλημα αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου περιφέρεια χρειάστηκε μόνη της να προκαταβάλει κάποια χρήματα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κάποια έργα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ρόλος των, των γαλλικών περιφερειών, γενικότερα των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λειτουργούν σαν τράπεζε και να προκαταβάλουν οι ίδιε ποσά, όταν αυτά πρέπει να προέρχονται κανονικά εξ αρχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια τραπεζίτες οι οποίοι χαίρονται ιδιαίτερα με την κατάσταση αυτή γιατί μπορούν και αποφελούνται. Θεωρώ λοιπόν γι' αυτό ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια κοινά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μας επιτρέψουν να έχουμε τη δική μας ταυτότητα απέναντι στις ε, μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των πρώτων υλών. Αν δεν καταφέρουμε να ασχοληθούμε με τον τομέα αυτό, φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε να καθυστερούμε πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χώρες, τρίτες ή αναδυόμενες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Είμαι πεπισμένος ότι από μόνες τους οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση εξατομικευμένα. Μόνο μέσω μιας συλλογικής κοινή δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Πρέπει λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει το δικό του το ρόλο. Εναπόκειται σε εμά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μιλήσουμε με πυγμή, με ιδιαίτερο σθένος, και θεωρώ ότι η συγγήτρια για το ζήτημα αυτό, όπως και για άλλα ζητήματα, έχει μιλήσει με ιδιαίτερα στεναρή φωνή και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε στο Συμβούλιο, να πούμε στο Συμβούλιο ότι ως εδώ και μη παρέκει, ότι ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον έχει άλλες απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και όλος ο κόσμος μας παρακολουθούν σε καθημερινή βάση. Όλοι περιμένουν να δούνε τι δράστα να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλά ζητήματα, όπως για το ζήτημα της ειρήνης για παράδειγμα, ή για το ζήτημα της Ουκρανίας, ή για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ή γενικότερα για την ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για όλους αυτούς τους τομείς να έχουμε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για να μπορούμε να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση. Από, τη, από τα ρωσοουκρανικά σύνορα μέχρι την γεωργική πολιτική, σε όλες αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των ε, γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν πλέον να εξαχθούν προς τη Ρωσία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και θα πρέπει, αν μη τι άλλο, τα προϊόντα αυτά, τα οποία δεν κατάφεραν να φτάσουν στη Ρωσία, να χρησιμοποιηθούν για την ανθρωπιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια γραμμή. Σας ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Ολμπράχτ. Ευχαριστώ. Απλώς να σας πω τις εξής παρατηρήσεις μου σήμερα. Έχουμε μια διτή συζήτηση, όπως πάντα όμως γίνεται με τον προπολογισμό κάθε χρόνο. Πρώτα-πρώτα η μία όψη είναι η τεχνική, η τεχνοκρατική όψη. Δηλαδή έχει, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και εμείς προτείνουμε οι εμπλεκόμενοι να δώσουν πράσινο φω για τα προγράμματα, αλλά δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να ε, προοικοδοτήσουμε αυτά τα προγράμματα. Να λοιπόν τι γίνεται. Έτσι γίνεται όταν λοιπόν ε, λείπουν χρήματα. Οι τοπικέ αρχέ, οι πάντες, οι πάντες ξέρουν ότι υπάρχει στενό της ρεύστου. Όμως η προκλήπη να λοιπόν, είναι ότι κάποιο όλα αυτά τα σχεδίασε ελπίζοντα ότι δεν θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Τα λέμε και ελπίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Αυτό είπανε, αυτό σκεφτήκανε. Ελπίζαν ότι όλα αυτά δεν θα ευοδοθούν και θα έχουμε και αναστολή κλπ. κλπ. Συγγνώμη που σας τα λέω έτσι ομά, αλλά έτσι γίνεται ο προγραμματισμός. Με την ελπίδα ότι δεν θα υλοποιήσουν. Όμως ευτυχώς γίνονται κάποια πράγματα γιατί η αποτελεσματικότητα είναι αποδοτικότητα, είναι καλύτερη από ό,τι πριν. Έχουμε αξιώσει ολένα και περισσότερε που σωρεύονται και θα πρέπει αυτέ να ικανοποιηθούν. Τη μία χρονιά μετά την άλλη μεταθέτουμε το πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Και ελπίζουμε ότι κάποιο κάποια μέρα θα το επιλύσει. Όμω, η άλλη όψη είναι η πολιτική. Ότι δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό-τεχνοκρατικό. Είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνώ με τους αδέλφους από το ECR. Από πλευράς των ευρωσκεπτικιστών η λογική λύση είναι περικόψατε πληρωμές ή περικόψατε τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Εντάξει, δεν συμφωνούμε, είμαστε ευρωσκεπτικιστές, είστε ευρωσκεπτικιστές και εμείς είμαστε φίλοι Ευρωπαίοι, χρειάζεται επομένω ένα μεγαλύτερος προπονός για μεγαλύτερη Ευρώπη. Εσεί θέλετε το αντίθετο. Λογικό αυτό. Όμω είναι πολιτικό το πρόβλημα. Εδώ θα το συζητήσουμε και θα βρούμε μια λογική λύση. Όμω το πρόβλημα είναι ότι το Συμβούλιο μην ξεχνούμε ότι η στρατηγική του 2020 φτιάχτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είπαμε τότε πόσο θα κοστίσει εμείς, πόσο θα κοστίσει η στρατηγική για το 2020 και είχαμε κάποιο είδους προσωρινό υπολογισμό και είπαμε δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για να εξυπηρετηθεί. Όμως συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Στρατηγική 2020. Έχουμε το πρόγραμμα. Όμως όλα τα κράτη-μέλη, όλοι και οι φιλευρωπαίοι και οι ευρωσκεπτικιστές συμφώνησαν. Και εμείς λέμε πού είναι τα χρήματα αυτά για να πέτυχουμε τους στόχους μας. Θέλετε οι στόχοι να καταπέσουν Θέλετε να υπάρξει περικοπή, λιγότερη Ευρώπη. Εμείς λέμε όχι, εσείς λέτε ναι. Δεν είναι αυτό τεχνικό, τεχνοκρατικό, είναι πολιτικό το πρόβλημα. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε το, το 3 και είχαμε αυτό το απόθυμα. Και τρία χρόνια μετά ε, κάνουμε αυτές τις διορθώσεις, Ελπίζω ότι κάποιος θα τα κάνει, γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Οπότε μην ε, λησμονείτε ότι είχαμε το πρόβλημα του πολιετούς, του δημοσιονομικού πλαισίου κλπ. Au fond, une Α, bon. Αυτά είναι καλά μαντάτα. Το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, φτιάχτηκε. Υπήρχε μια διαφορά μεταξύ των πιστώσεων πληρωμών και πιστώσεων υποχρεώσεων και αφετηρία ήταν η αρχή ότι, όλα αυτά δεν θα υλοποιηθούν γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα ούτως ώστε αυτοί που ανέλαβαν να μπορούν να υλοποιήσουν και να τρέξουν τα προγράμματα. Όμως τα καλά τα σήμερα ποια είναι ότι τα προγράμματα αυτά λαμβάνουν σάρκα και οστά και επομένως θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα και θα πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε πιο συνεπείς όσον αφορά την εξισορρόπηση πιστώσεων πληρωμών και πιστώσεων υποχρεώσεων. Ε, αν κανείς δεν είναι αισιόδοξο, δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική. Έτσι είμαστε κι εμείς, αλλά είναι και θέμα τώρα μέτρου. Ίσως η Επιτροπή μας καθησυχάζει όσον αφορά ε, το που καταλήγουν και με τη χρονοδιάγραμμα εξελίσσονται οι υποχρεώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι σωρεύει υποχρεώσεις, σωρεύει οφειλές, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Όλο και περισσότερο, αλλά πριν δώσω το λόγο στην κυρία Καλβίνο, θέλει το λόγο κύριο Ζανίου. Μάλιστα. Είχα προηγούμενα ζητήσει να μπορέσω να παρέμβω. Αλλά σε σχέση με το, τις εργασίες εδώ, μάλλον με αγνοήσατε, θα προσπαθήσω να συνοψίσω γιατί πολλά αναφέρθηκαν. Πρώτα ευχαριστώ την εισηγήτρια για την διεξοδική και περιεκτική και εξαντλική παρουσίαση των στόχων. Ακόμα και αν μια πρώτη ανάλυση των θέσεων του Συμβουλίου μόνο τότε μπορεί να γίνει και να επιτευχθεί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά την πολιτική των κρατών μελών θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει όταν εδώ υπάρχουν τα θέματα περικοπών και εξοικονόμησης κονδυλίων είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πορεύεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αν όμως αναλύσουμε την πρόταση του Συμβουλίου τότε βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις βλέπουμε συγκεκριμένα ότι γίνονται ορισμένες προτάσεις οριζοντίων περικοπών χωρίς να γίνεται μια συγκεκριμένη ανάλυση των επιπτώσεων των περικοπών αυτών, των επιπτώσεων που θα έχουν δηλαδή για τον κοινοτικό προπολογισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξορθολογήσουμε τους πόρους, σίγουρα, αλλά από την άλλη, παράλληλα, θα πρέπει ο κοινοτικός προπολογισμός να επικεντρωθεί στις πραγματικές προτεραιότητες, τις οποίες ακούσαμε από τους ε, ευρωβουλευτές από τον ίδιο τον, πρόεδρο της, ε, τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται για προτεραιότητες ε, που έχουν εγκρίνει ακόμα και οι ίδιοι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε για τις πολιτικές εκείνες που υποστηρίζουν την απασχόληση, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι πολιτικέ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερο τη βιομηχανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε επίση χρηματοδοτικά και τι πολιτικέ για την έρευνα. Η έρευνα αποτελεί μια σημαντικότατη βάση για την οικονομική ανάπτυξη. Χωρί έρευνα δεν υφίσταται πρόοδο, δεν υφίσταται εξέλιξη, δεν υφίσταται οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση για την περικοπή των πληρωμών. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι, αποτελεί όνειδος η πρόταση του Συμβουλίου το Συμβούλιο με ένα παράδεκτο τρόπο προσεγγίζει το ζήτημα αυτό και από ό,τι φαίνεται δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, όπως είπε και η σοσιαλίστρα συνάδελφος, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάθε χρόνο χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες πτωχεύουν, οι οποίες καταστρέφονται. Το έχουμε δει αυτό πολύ έντονα στη χώρα μου, την Ιταλία. Και πτωχεύουν οι επιχειρήσεις αυτές όχι επειδή δανειοδοτήθηκαν με υπερβολικά ποσά, όχι επειδή δεν λειτουργούν σωστά ή δεν υποβάλλουν σωστές υπηρεσίες, αλλά γιατί δεν καταφέρουν να κτίσουν τα χρήματα εκείνα τα οποία τους οφείλονται. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός αυτό. Θα πρέπει να καταφέρουμε να μειώσουμε το τεράστιο αυτό χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών και θεωρώ ότι η υποχρέωση που έχουμε ως Επιτροπή Προεπολογισμών απέναντι στο Συμβούλιο είναι να δείξουμε μία στεναρή στάση και να καταφέρουμε να πείσουμε το Συμβούλιο ποιε είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από τις προτάσεις οποίες έχει υποβάλει. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Καλβίνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α είστε σύντομοι σα παρακαλώ πολύ γιατί έχουμε ακόμα πολλά σημεία στη μερίσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα, γενικά, μια παρατήρηση για αυτά που συζητάμε και μετά θα αναφερθώ στο θέμα του γέστα λικίντε των υπολείπων προς εξόφληση που αναφέρθηκαν. Πρώτον, η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες της, ε, της εισηγήτριας για τον πολύ περιοριστικό, την πολύ περιοριστική αντιμετώπιση από βράση του Συμβουλίου και επίσης συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις που έγιναν για την αντίφαση μεταξύ της θέσης του Συμβουλίου και των πολιτικών δηλώσεων που έχουν γίνει. Θεωρητικά θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες σε εκείνες τις προτεραιότητες που δίνουν αύξηση στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Στην πρακτική όμως, αν δούμε σωστά την θέση του Συμβουλίου, η κατηγορία 1α είναι μια αρνητική προτεραιότητα πλέον. Γι' αυτό συμφωνούμε απόλυτα με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σήμερα. Η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι η εξής. Τονίζει επίσης ε, και εντάσσεται και σε άλλες παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών σήμερα λέγοντας ότι υπάρχει υποχρέωση να υπάρχουν επαρκείς πληρωμές ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις πληρωμών. Προηγούμενες δηλαδή υποχρεώσει που έχει υπογράψει το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, τα θεσμικά όργανα. Και είναι σαφή και διαφανή η συνθήκη και στο άρθρο 323 όταν λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα διασφαλίζουν ότι τα δημοσιονομικά κοινά μέσα θα διασφαλίζονται ώστε να μπορέσει τι νομικέ υποχρεώσει να τι αντιμετωπίσει έναντι τρίτων ε, συμβαλωμένων μερών ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν μια συνθήκη που θέτει σαφώ τι υποχρεώσει. Και είναι σαφέ και πρέπει να τονίσουμε ότι αναφερόμαστε σε προηγούμενε υποχρεώσει που έχουν αναλυφθεί και δεν είναι καθόλου τεχνική αυτή η συζήτηση όπως αναφέρθηκε. Υπάρχει εδώ μια ανισότητα πληρωμών σε σχέση με τις υποχρεώσεις. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Οι παλαιές υποχρεώσεις πρέπει να εκτελεστούν. Και αν δεν υπάρξει προσυπογραφή και εκτέλεση των υποχρεώσεων για προγράμματα τα οποία πρέπει να εκτελεστούν, δεν θα υπάρξει υλοποίηση των πολιτικών μας. Αυτά που συζητάμε είναι για μια πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Δηλαδή θα υλοποιηθούν τα μέσα για την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί ή όχι. Δεν είναι μια τεχνική φύση συζήτηση. Εδώ υπάρχει κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί μέσω αυτών των δράσεων. Και τρίτον, και απορρέει από αυτά τα οποία προανέφερα, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν, να δούμε το θέμα δημιουργίας ρεαλιστικών περιθωρίων. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, καταλήγουμε σε διορθωτικούς προϋπολογισμούς με δραματικά αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε επαρκή κονδύλια, θα έχουμε σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών και κάθε φορά θα έχουμε μια τέτοια συζήτηση και οι πολίτες θα θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί διαρκώς νέα κονδύλια ενώ εμείς είχαμε πει ευθύς εξ αρχής ότι απαιτούνται αυτά τα κονδύλια ευθύς εξ αρχής για να υλοποιηθούν υποχρεώσεις που έχουμε υπομειστεί. Τώρα, για το θέμα των υπόλοιπων προς εκτέλεση και κάποια άλλα συναφή τα οποία προαναφέρθηκαν σήμερα, δύο τρίτα των υπόλοιπων αυτών αφορούν την πολιτική συνοχής και αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν αρκετά δύσκολο να προβλέψει κανείς εξειδικευμένα πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά, διότι εξαρτώνται από την υλοποίηση των προγραμμάτων το γεγονό ότι υπάρχει αύξηση των υπολείπων προ εξόφληση είναι φυσιολογικό αν λάβουμε υπόψη την αύξηση, σαφή αύξηση, διαρκή αύξηση των ε, υποχρεώσεων μέχρι το 2013. Αλλά όπω εμεί λέγαμε με κάθε συνέπεια αυτό το κενό μπορεί να αντιμετωπιστεί αν τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια μπορέσουν να υλοποιηθούν πλήρω και έχουμε και τα πλαίσια ελαστικότητα τα οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν σε σχέση με την υλοποίηση των πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο για τις ε, πληρωμές για το 2015. Γι' αυτό προτείναμε στο σχέδιο προϋπολογισμού 2015 την εκτέλεση του 100% του ε, περιθωρίου των ε, δυνατοτήτων για τις πληρωμές. Για τα πιλωτικά προγράμματα, πολύ σύντομα, να πούμε ότι μας ικανοποιεί το πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση τώρα με παρατηρήσεις που έγιναν δεν τις δεχόμαστε εργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο θετικά και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει η βέλτιστη εφαρμογή δημοσιονομικά όλων αυτών των προγραμμάτων γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί και όπως ανέφερε και η ίδια η συγγήτρια αλλά επιτρέψτε να δώσω ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα να πω ποιε είναι οι επιπτώσει ή ποιε είναι οι αντιφάσει σε σχέση με τι πιστώσει πληρωμών. Αρκετοί από εσά ανέφεραν το πιο, την πιο προφανή αντίφαση με την κατηγορία 1α και την κατηγορία 4. βλέποντα εξειδικευμένα τη θέση του Συμβουλίου, ένα σαφέ παράδειγμα είναι η έρευνα. Αρκετοί από εσά αναφερθήκατε στην έρευνα. Εκεί υπήρξε περικοπή στα κονδύλια για το ε, πρόγραμμα, το 7 πρόγραμμα για την έρευνα. Δηλαδή δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν κονδύλια και θα υπάρξουν καθυστερήσεις και θα πρέπει να υπάρξει μετάθεση εκτέλεση εκτέλεσης αυτών στον επόμενο προϋπολογισμό του επομένου έτους. Αν δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες υπάρχουν σαφείς επιβαρύνσεις και επιπτώσεις. Και ένα δεύτερο επίπεδο ασαφίας και ε, αναντιστοιχίας είναι σε σχέση με τα όσα γίνονται στην γειτονιά γωνιά της ε, Ευρώπης και των προβλημάτων που αυξάνονται τα προβλήματα και υπάρχουν περικοπές στα κονδύλια σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού. Δύο παραδείγματα για το μίσο του όπου υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Ετσενικέ ήθελε να πάρει τον λόγο. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι γνώσει μου για τον προπολογισμό είναι στοιχειώδε. Όμως, έχουμε εδώ πέρα κάποια θέματα γενικότερα για τα οποία μπορώ να σχολιάσω. Πρώτα-πρώτα, έχουμε την Τρόικα, η οποία τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση τις εκβιάζει. Είναι θέμα των χρεών, όπως το των πολύ η Ένωση είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την σόρευση των οφειλών της. Έχουμε επομένω αυτό το, το, το, το, το παιχνίδι του, του καλού μπάτσου και του κακού μπάτσου. Και έχουμε 1,5 δις και, το, και τη σχετική οροφή που έχει τεθεί από το πολιετές πλαίσιο. Ζητάμε και τις, έχουμε και αυτές τις περικοπές των 500 εκατομμυρίων παραπάνω. Ελπίζω ότι υπάρχει συνένεση για το ότι θα πρέπει οι πιστώσεις να διατεθούν ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις οφειλές μας και μην έχουμε μόνο περικοπή των πιστώσεων. Merci. Euh, Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ε, Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και είδα μεγάλη απόκληση απόψεων βέβαια. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα χρέους, το οποίο συνεχώς διωγγώνεται. Πρόκειται για ένα τεράστιο χρέος, επιζήμιο, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο αντιβαίνει στο πνεύμα της συνθήκης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δανείζεται και υπερχρεώνεται, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τη συνθήκη, άρα πρέπει να βρούμε γι' αυτό μια λύση σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Και όσον αφορά το μέλλον, σίγουρα δεδομένου το ότι τα κράτη-μέλη θα θέλουν να υλοποιούν τα προγράμματα τα οποία έχουν εγκρίνει και δεδομένου ότι θα θέλουν να χρησιμοποιούν το τμήμα του προπολογισμού το οποίο προβλέπεται για αυτά, θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τόσο τεράστια περιθώρια στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να προβλέψουμε για περίοδο επταετίας τι μπορεί να συμβεί. Ξέρετε πόσο ευμετάβλητη είναι αυτή τη στιγμή η οικονομία, πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να ανταποκρίνεται περισσότερο στην επικαιρότητα, δηλαδή στα όσα προκύπτουν την τελευταία στιγμή, στα όσα προκύπτουν συγκυριακά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρει και η συγκήτριά μας να καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα μετά τη συζήτηση αυτή και ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να μας βοηθήσει στην πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που θα έχουμε με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Γκαρθιά Σαμπάλ, έχετε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Η συγκήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, αλλά βέβαια και εγώ ως εισηγήτρια δεν μπορώ να επιτελέσω αυτό το έργο μόνοι. Θα προσπαθήσω να συγκεράσω τις επιμέρους θέσεις του Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε από ό,τι άκουσα για το πώς αναλύουμε την κατάσταση και σε σχέση επίσης ε, τώρα συμφωνούμε με, με, με, το που θέλουμε να καταλήξουμε για μην συμφωνούμε τόσο πολύ με τη μέθοδο για άκουσα και τον κύριο Άλμπριχτ ότι δηλαδή ε, είμαστε από τη μία μεριά οι φιλοευρωπαίοι ε, και την άλλη μεριά οι ευρωσκεπτικιστέ. και επομένως ισχύει ότι ο προπολογισμό είναι αφορμή περισκέψη προβληματισμού για το πώς βλέπουμε από πολιτικής πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν πραγματικά είμαστε φιλευρωπαίοι και αν θεωρούμε ότι είναι ένα όραμα αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να το προχωρήσουμε αυτό το όραμα. Από πλευρά προπολογισμού είναι καλύτερα να έχουμε τέτοια κοινά προγράμματα με προ... κοινέ ε, ε, Αυτό είναι ένα τρόπο, μια μέθοδο ε, ε, διευθέτηση του προπολογισμού. Τότε, τότε υπάρχει πραγματικά προτιθέμενη αξία. Αλλιώς, τι να εξυπηρετήσει άλλο ο προϋπολογισμός. Γι' αυτό και πέραν του αν θα έχουμε ή όχι περικοπές, αλλιώς δεν θα τον προπολογισμό, σας τον καταργούσαμε. Επομένως, ακριβώς χρειάζεται και γι' αυτό θα πρέπει να τον αυξήσουν τον προπολισμό, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να τον αυξήσουμε βελτιώνονται τα προγράμματα, βελτιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης έτσι εξοικονομούν χρήματα και τα κράτη-μέλη. Άρα ανάλογα επομένω με το πώς από πολιτική πλευρά βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και υιοθετούμε την ΑΒ θέση για τον προπολογισμό επίσης. Μου άρεσε αυτά που είπε η κυρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πάρα πολύ σαφής όσον αφορά ε, τις εξηγήσει και ε, κάποιο είδους ε, άλλα δεδομένα τα οποία είπε που είναι σημαντικά, ας πούμε η βοήθεια μας, η βοήθεια αυτή που μας δίνει τέλος πάντων είναι πάρα πολύ σημαντική ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματούμε το Συμβούλιο και να μπορούμε να γνωρίζουμε ε, πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχουν οι υπολογισμοί και ακούσαμε πολλά για το ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας Κανείς, κανείς από όσους μίλησαν δεν είπε κάτι αντίθετο. Όμως, να γίνει εδώ μια διάκριση. Πρώτα-πρώτα έχουμε κάποια προγράμματα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και ε, εκεί εκκρεμούν κάποια χρέη. Αυτό δεν είναι καν ε, υποχρέωση. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Είναι γεγονός. Υπάρχουν πόλεις, υπάρχουν περιφέρειες, προγράμματα περιφερειακά, εκεί που έχουν προκαταβάλει χρήματα εκείνη, τα οποία δεν τους έχουν καταβληθεί. Δεν πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχουν όμως και διάφοροι, διάφορες υποχρεώσεις από την άλλη μεριά που προβλέπονται από το πολίτες πλαίσιο και όλα αυτά είχαν προγραμματιστεί και έγινε αυτός ο προγραμματισμός για όλα τα προγράμματα Επομένω αυτά τα οποία προγραμματίστηκαν θα πρέπει να τα τηρήσουμε και πρόκειται επομένω για όλου αυτού οι οποίοι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βάσει αυτού του είδου τον οικονομικό προγραμματισμό, τον προσωρινό προγραμματισμό. Ε, όλα αυτά είναι δεσμεύσει που θα πρέπει να τηρηθούν. Δεν μπορούμε εκεί να περικόψουμε τίποτα. Θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Και με αυτά τα προβλήματα Είδα ότι έχουμε εδώ τις δύο κατηγορίες, τις δύο στήλε, υποχρεώσεις, πληρωμές. Τι μου είπανε στην αρχή. Στην αρχή μου είπανε μην, μην, μην, ε, μην κουράζεσαι για τις πληρωμές, ασχολήσουμε με τις υποχρεώσεις. Ενά που δεν είναι έτσι τα πράγματα που τώρα ακριβώς κατέστησαν οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις το ίδιο σημαντικά. Άρα θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα γίνει, πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ορισμένες ε, επενδύσεις που έχουν στατική σημασία για το μέλλον. Έχουμε όλα αυτά τα οποία λέμε ότι θα πρέπει να πληρωθούν. Τα καθημερινά έξοδα είναι δυνατόν, είναι απίστευτο ένα θεσμικό όργανο να μην πληρώνει τις οφείλες του. Πέραν του εδώ είπαμε ότι έχουμε ε, φιλοευρωπαίους προσκεπτικιστέ, η δική μου δουλειά ως συγκίτρια είναι να, τα, να συγκιάζω αυτές τις απόψεις και να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να μας ε, αναδείξει σε ισχυρού συνομιλητέ στις διαπραγματεύσει. Οπότε, θα επεξεργαστούμε τις ε, τροπολογίες των ε, ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών θα κάνουμε συναντήσεις με πολιτικές ομάδες, με συναδέλφους και θα καταλήξουμε έτσι σε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Χολμαϊρ, θέλετε να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε τα άλλα κεφάλαια, τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού μέσα σε αυτό το στενό χρονικό πλαίσιο. Μα έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω εργασία ε, οι διερμηνεί και του ευχαριστούμε. Έχουμε του προσκεκλημένου, τον εκπρόσωπο επίση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να δούμε τι θα γίνει με τι επενδύσει. Τι μπορεί να γίνει ούτω ώστε να προχωρήσουμε προ τα εκεί καλά. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να είμαστε σύντομοι. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε μια διορθωτική επιστολή που θα λάβουμε. Τότε θα έχει νόημα να συζητήσουμε τον προϋπολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι σήμερα που δεν έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Δεύτερο, αυτό το οποίο σε σχέση με την Επιτροπή, τον προϋπολισμό της Επιτροπής συζητήσαμε, αφορά και τον προϋπολισμό των άλλων τμήματων. Δηλαδή έχουμε δύο ξεχωριστά προβλήματα εδώ που δεν ασχολήθηκε το ίδιο το Συμβούλιο. Και έχουμε το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει έναν δεύτερο γενικό εισαγγελέα και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αναγκαίες θέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η δεύτερη εισαγγελική θέση έχουν περικοπεί. Και αυτό Στη συνέχεια, δεύτερο, το Συμβούλιο αύξησε το ποσοστό, όμως δεν πρόσεξε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με μια επιβάρυνση 99% σε σχέση με το προσωπικό επιβαρύνεται. Αν δούμε τώρα το ποσοστό, το οποίο σε σχέση με το δικαστήριο αυξάνεται, ενώ δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο αύξησης, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να ε, στελεχωθούν αυτές οι θέσεις. Και έχουμε το 48, το, την προθεσμία 48 ε, ε, μήνων που δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Προβλήματα που δημοσιονομικά μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Έχουμε την πρώτη προσφυγή μιας επιχείρησης για 13 εκατομμύρια ζημιά που έχει υποστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή η υπόθεση αυτή εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε και άλλες τέσσερις προσφυγές οι οποίες ε, συνεπάγονται πολύ μεγαλύτερα κονδύλια διότι πρόκειται για δισεκατομμύρια απαιτήσεων. Αυτά όλα τι σημαίνουν σαν συνέπεια. Μια και το Συμβούλιο είχε πει ότι οι πρόσθετοι δικαστές ε, θα έπρεπε να αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εννέα τουλάχιστον κατά τον αριθμό, όμως εδώ και 1,5 χρόνια, 1,5 χρόνο δεν υπάρχει συμφωνία πώς, από ποιες χώρες θα στελεχωθούν διότι 28 χώρες ε, αν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν έτσι και έχουμε πρόβλημα για αυτές τις 9 θέσεις δικαστών και δεν μπορούν να στελεχωθούν υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να στελεχωθούν αυτές οι θέσεις 9 δικαστών αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τον επιμερισμό από ποιε χώρες θα στελεχωθούν. Είναι μια φάρσα αυτό και αυτό μπορεί να έχει τεράστιες δημοσιονομικές επιπτώσεις βάρος μας δημοσιονομικά. Γι' αυτό το λόγο από πλευράς μας θα ήθελα να παρακαλέσω την ε, Επιτροπή μας ε, για το ε, Ευρωπαϊκό, Δικαστήριο πρώτον να αναμείνουμε τις προτάσεις να αποσυρθούν οι προτάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως έχει προταθεί διότι διαφορετικά θα έχει σημαντικότατες επιπτώσεις βάρος του προϋπολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η κατάσταση. Όταν θα, αν, κερδίσουν αυτές τις προσφυγές αυτές οι εταιρείε, τότε θα υπάρξει απέτηση επιστροφής κονδυλίων ε, και αν δεν ε, κερδίσουν αυτή την προσφυγή τους ε, τότε θα έχουμε επιβάρυνση σε σχέση με τον προϋπολογισμό μας λόγω προστήμων και στις δύο περιπτώσεις θα επιβαρυνθούμε. Δεν δείχνουμε λοιπόν καμιά κατανόηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για το πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή και το Συμβούλιο αυτό το πρόβλημα η νομολογία θα πρέπει μέσα σε ένα αποτελεσματικό χρονικό διάστημα να μπορεί να επιτυγχάνεται από πλευράς αποφάσεων δικαστηρίων, δικαστηρίου και θα πρέπει λοιπόν λόγω της, της εύλογης χρονικής ε, διάρκειας ε, ε, των αποφάσεων αυτών να δράσουμε. Γι' αυτό θα προετοιμάσω τροπολογίες ώστε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να υπάρξει υποστήριξη που θα διασφαλιστεί ώστε για το ελάχιστο αναγκαίο να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτές τις θέσεις στο ελάχιστο το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι το Συμβούλιο επιθυμεί να μην υπάρχει, να, ε, να είχε ε, εξαλειφθεί η υπηρεσία υπηρεσία, η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Αρχικά υπήρχαν συμφωνίες από το Συμβούλιο και είχε πει το Συμβούλιο ότι θα διασφάλιζε τη στελέχωση και την χρηματοδότηση. Μετά την επόμενη χρονιά είπαν ότι όχι, δεν θα το κάνουν αυτό θα έπρεπε να ε, αναλάβει την ίδια την ε, ε, ευθύνη το Συμβούλιο. Και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε μόνο θεσμούς IT που θα μέσα στο YouTube μεταξύ κυρίας Άστον και τον ε, ε, ποιος ήταν ο τελευταίος ο Υπουργός Εξωτερικών της Εστονίας νομίζω ήταν ή της Λετωνίας αλλά όλα αυτά μπορεί να τα δει κανείς στο YouTube πως τηλεφωνούσαν και τι ήταν το, ποιο ήταν το αντικείμενο των συμφωνιών και των συνδιαλέξεων αυτό μπορεί κανείς σε σχέση με τους ε, εξωτερικούς ε, ε, αντιπροσώπους που έχουμε να το κάνει κανείς. Έχουμε ένα ανεδαφικό παλαιό πρόγραμμα το οποίο ένας απλός hacker μπορεί να προσβάλλει και να αντλήσει στοιχεία από αυτό και δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια. Και θα έπρεπε να δούμε ότι από το 1998 υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο ασφάλειας. Με τα σημερινά προγράμματα ε, κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο να αποκαλύπτονται τα στοιχεία ε, σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, τότε λοιπόν βλέπουμε τι συμβαίνει με την περικοπή και διαγραφή των κονδυλίων σε σχέση με την εξωτερική υπηρεσία. Αυτή είναι η κατάσταση. Καμιά φορά τα πράγματα είναι όπως στο νηπιαγωγείο. Υπάρχουν ε, θέματα τα οποία είναι πολύ εύληπτα, δεν είναι καθόλου δύσκολα να τα κατανοήσει κανείς και ουσιαστικά θα έπρεπε με την κοινωνική, κοιν, κοινή λογική να μπορούν να ρυθμιστούν. Αλλά όμως δεν ρυθμίζονται. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επεκταθώ περισσότερο στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στον προϋπολογισμό μας, για τον προϋπολογισμό τους όταν θα έχουμε τη διορθωτική επιστολή θα μπορέσει να διασφαλιστεί η αντιστάθμιση διότι έτσι θα μπορέσει να υπάρξει αποτελεσματικότητα για τον προϋπολογισμό που σε δύο εβδομάδες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα και να τα διευθετήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να προσθέσω εκτός από αυτές τις δύο παρατηρήσεις. Merci, ευχαριστούμε κυρία Χολμάιερ. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε μια ολόκληρη συζήτηση, διότι ε, πρέπει να μιλήσουμε και για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τα ομόλογα έργου. Αν δεν υπάρχει κάποια επίγουσα ερώτηση για τα όσα είπε η κυρία Χολμάιερ, να την ευχαριστήσουμε τη συνάδελφό μας, επειδή πραγματικά τόνισε τα προβλήματα τα οποία υφίστανται όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάδει με την ε, ενιαία αγορά. Ενιαία αγορά σημαίνει θεμητός ανταγωνισμός. Αν λοιπόν χρειάζονται να περάσουν πάρα πολλοί μήνες προκειμένου να εκδικαστούν υποθέσεις στο δικαστήριο που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, τότε αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει οτιδήποτε κακό κείμενο δηλαδή μπορεί να συμβαίνει στην εσωτερική μας αγορά και αυτό επηρεάζει προφανώς την οικονομία μας, την ανάπτυξη αλλά ακόμα και τις θέσεις απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τα πρόστιμα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να εγγραφούν στον κοινοτικό προπολογισμό και τα οποία καθυστερούν ακριβώς επειδή δεν εκδικάζονται γρήγορα υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας καλώ λοιπόν κύριε Χολμάιρ να λάβετε δράση προκειμένου να ταρακουνήσετε λίγο το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει, παρακαλώ. Είναι πραγματικά σκανδαλώδε το ότι πρέπει να περάσουν 48 μήνες για να εκδικάσουμε υποθέσεις. Δεν λειτουργεί, δυσλειτουργεί η ενιαία αγορά μα. Συμφωνώ, συμφωνώ 100% κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπατε για την καθυστέρηση αυτή. Θα ήθελα μόνο να πάρω το λόγο πολύ σύντομα για να σας εξηγήσω ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν έχει ως στόχο να μειώσει τους πόρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το αντίθετο μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας ε, την αύξηση των ε, πληρωμών που πρέπει να έχουμε για τη νέα θέση Γενικού Εισαγγελέα Προσπαθήσαμε όμως οριζόντια να εφαρμόσουμε μία μείωση 5% στο προσωπικό, η οποία ξέρετε ότι έχει επιβληθεί σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε το θετικό παράδειγμα και μάλιστα μειώσαμε πάρα πολύ το προσωπικό μας το τελευταίο διάστημα και μειώσαμε κατά συνέπεια και τις σχετικές δαπάνες στον προπολογισμό μας και προσπαθήσαμε να έχουμε μία συνεπή στάση και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Αναφερθήκατε βέβαια σε δύο, τα οποία ουσιαστικά παρουσιάζουν αυξήσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Τονίζω πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σε καμία περίπτωση περιοριστική προσέγγιση προσπαθεί απλώς να πετύχει μια συνέπεια, μια συνεκτικότητα στη στάση που κρατάνε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πρόεδρος γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα και ότι όντως λαμβάνονται αποφάσεις οριζόντιες τις οποίες πρέπει να τηρήσουν όλα τα θεσμικά όργανα. Πολλές φορές όμως προκύπτουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σωστές, δεν είναι θετικές και καλούνται οι πολιτικοί να διορθώσουν τα κακό κείμενα. Κυρία Χολμάιερ, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση στο σημείο αυτό για τα τμήματα του προπολογισμού που μας παρουσιάσατε. Θα περιμένουμε τώρα λίγο τους ε, προσκεκλισμένους μας όσον αφορά τα project bonds. Ο κύριος Γκόραν Φάρμα, ο προηγούμενος συγητής μας για το ζήτημα αυτό, δεν είναι πλέον μέλος της Επιτροπής μας. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Τζόρτζιο Κασόνη, επικεφαλής της ΕΚΦΗΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι επικεφαλής για τις πολιτικές υποδομών, και στον Νάιτζελ Τζάνετ, ο οποίος είναι διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όσον αφορά κάποια νέα προϊόντα και κάποιες ειδικέ συναλλαγές. Κύριοι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε να παρουσιάσουν αυτή την έκθεση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας συνοψίσουμε την κατάσταση. Πώς δηλαδή έχουν τα πράγματα σήμερα για αυτά τα ομολογιακά δάνεια. Πάρα πολύ δραστήρια στάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κατάτμιση αυτών των ε, υποστηρίξει αυτών των, των επενδύσεων, ούτω ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Έχουν γίνει πάρα πολλά συνεργασίε, αλλά ακόμα έχουμε έργο μπροστά μα. Το Μάρτιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προέβη στη σχετική ανακοίνωση για το τι θα χρηματοδοτήσει για αυτές τις δράσεις, ε, για το τι προβλέπεται. Τώρα, Από πλευρά ζήτηση έχουμε πολλά να κάνουμε. Ο κ. Γιούνκερ αναφέρθηκε σε αυτά τα 300 δις. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τις λεπτομέρειες αυτών των κατευθυντηρίων που περιέγραψε ο κύριος ε, Γιούνκερ. Σε επίπεδο όσα και G20 συζητείται η υπόθεση. Και τώρα, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε το πιο σωστό πλαίσιο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στους δύο βασικούς τομείς εκεί που θεωρήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, δηλαδή μήμη ε και υποδομές. Επομένως θέλουμε αυτά τα ομόλογα τώρα να υποστήξουν και τα έργα και προγράμματα υποδομής. Για να σας ε, υπενθυμίσουμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση με αυτά τα μολυγιακά δάνεια. Χρειάζονται επενδύσεις, είπαμε, για κάποια προγράμματα ενός 3 με το 2020 που έχουν σχέση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Βεβαίως και υπάρχουν ε, τα προβλήματα στενότητα των εθνικών προπολογισμών και άρα ε, περισσότερο τώρα θα πρέπει να προσφύγουμε στον ιδιωτικό τομέα για να χρηματοδοτηθούν αυτέ οι επενδύσει. Στα πλαίσια αυτά, αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012. Ε, Ευτυχώ το υπεστήριξε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξεκίνησε το 2012. 2013 Είχαμε ε, την πρώτη συμφωνία που επετεύχθη και έγινε ε, αυτή η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης το καλοκαίρι. Και έχουμε τώρα για τα ομολογικά αυτά δάνεια για αυτές τις εκθέσεις για τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα προς το Κοινοβούλιο. Και έχουμε αυτή την ενδελεχή έκθεση, αυτή η οποία ολοκληρώθηκε. Οπότε, αυτό το οποίο θέλαμε είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κεφαλαιοχικέ ε, επενδύσει, γιατί είχαμε μακροπρόθεσμε περικοπές που αφορούσαν αυτά τα, τα δάνεια, τα μακροπρόθεσμα, άρα θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε τα, τους σχετικούς πόρους από διάφορα θεσμικά όργανα, ούτω ώστε οι επενδυτέ να στραφούν προς τα εκεί που θέλαμε. Και επίσης θέλαμε ε, το νοηγητικό και το παθητικό να έχουν κάποια αντιστοιχεία, ας πούμε ε, υποδομές, ας πούμε άλλο, άλλο, άλλες υποχρεώσεις να είναι έτσι η ισορροπία τους, ούτως ώστε προς αυτές τις πρωτοβουλίες να στραφούν ευχαρίστως οι επενδυτές. Μέχρι σήμερα έχουμε κλείσει πέντε τέτοιες συναλλαγές σύμφωνα με αυτή την πρωτοβουλία μουλιακών δανείων για το νέο προπολογισμό και σε αυτή την φάση έχουμε την προϋποδότηση 230 εκατομμυρίων για κάποια προγράμματα τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν μέχρι το τέλος του 2014 και να φτάσουν μέχρι το 2016 και είπαμε τουλάχιστον για τα πρώτα δύο χρόνια σύμφωνα με το Connecting Europe προχωρήσουμε, να 2015 να έχουμε μια αξιολόγηση και να αποφασιστεί το τι θα γίνει, ε, πώς θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία και αν θα συνεχιστεί. Ο συνάδελφος δίπλα μου θα σας πει πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με τα επιμέρους προγράμματα, αυτά τα οποία υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία, αλλά σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μόχλευση από τον προϋπολογισμό και έχουμε τα υπόλοιπα αυτών των 230 εκατομμυρίων τα οποία πρόκειται να πάνε στο, στο καταπίστευμα για το λογαριασμό αυτών που αφορά τα μολογικά δάνεια και όσον αφορά το, έχουμε, το συνελ, έχουμε 4 δις μέχρι το 2030 οπότε και θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τη μόχλευση αυτά τα ε, δάνεια ούτως ώστε να έχουμε ένα μαξιλαράκι ούτως υπήν όσον αφορά την, αγορά αυτών των δανείων από τους εξωτερικούς ε, ε, επενδυτές. Δεν είναι πλήρης η κάλυψη, απλώς υπάρχει για την πρώτη δόση ε, μία κάποια πίστοση. Τώρα, εμείς επομένως δεν, δεν 100% της έκθεσης, αλλά περίπου 30% της ε, έκθεσης της ΕΤΕ για αυτές τις ε, συναλλαγές, transactions. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι από το 2007 ε, υπάρχει μια μεγάλη μείωση των ποιοτικών επενδύσεων στην υποδομή. από το 2007 μέχρι το 2013 έχουμε πέσει σχεδόν κατά 50% και αντίστοιχα επίσης από το 2007 PPP μειώθηκαν κατά 30% και είναι αυτού του είδους τα, τα προγράμματα τα που χρηματοδοτεί ο ιδιωτικός τομέας. PPP συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου. Και οπότε έχουμε και αυτά τα δάνεια για τις υπόλοιπες δραστηριότητε είναι αλήθεια ότι υπάρχει για την ε, ταμιακή ροή πρόβλημα, υπάρχει στενότητα. έχουν τα stress test τα οποία ακριβώς έχουν ε, στριμώξει τις τράπεζες. Ε, και οι τράπεζες θα είπαμε ότι σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό που ισχύει τώρα θα δανείζουν όλο και περισσότερο βράχη πρόθεσμα. Τώρα, εδώ είναι το μεγάλο, το, μεγάλο μειονέκτημα δύνατο σημείο είναι ότι παρά το ότι υπάρχει πρόθεση θετική από τους επενδυτές αλλά υπάρχει πρόβλημα με την ζήτηση. Δεν είναι έτοιμα, δεν είναι όριμα κάποια προγράμματα που πολύ λίγα φτάνουν στην αγορά, είναι πάρα πολύ άγριος ο ανταγωνισμός οπότε αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει η προσοχή μας στο, στο πού χρειάζεται η υποστήριξη και να δούμε πού υπάρχει ε, καλή πλαισίωση από, τις, ε, από την αρχή, τη δημοσία αρχή η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα. Ε, τώρα έχουμε κάποιες ε, και σε διαφάνειε, δεν έχουμε μεγάλη σημασία. Πάμε παρακάτω. Να δούμε επίσης πόσο έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα. Έχουμε τέσσερις ε, ε, δράσεις και συναλλαγές που υποστηρίζουν τον πολιτισμό εξωτερικοί διαγωνισμοί, ε, αυτή η πρωτοβουλία θεωρείται ότι χτίζει, βοηθάει την αγορά. Η, η τράπεζα υποστηρίζει, δίνει αξιοπιστία στην αγορά. Πάντως, θα σας πει ο συνάδελφος ότι θα τηρήσουμε, θα πετύχουμε το στόχο μας για τα 5 έως 7 ε, προγράμματα. Είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία από τα προγράμματα τα κυβερνητικά. να αρθούν οι αβεβαιότητες σε σχέση με το τι κάνουν οι αρχές όσον αφορά αυτά τα ε, δάνεια. δεν είναι μια εύκολη λύση, μια εύκολη μέθοδος αυτά τα δάνεια, αλλά θέλουμε να επεκταθεί η χρήση όχι μόνο σε χώρες υψηλής αξιολόγησης που είναι εύκολα αλλά και σε κάποιες χώρες χαμηλότερες αξιολόγησης. Αυτό θα είναι η επόμενη φάση της πρωτοβουλίας και τώρα. Για την Connecting Europe Facility είπαμε ότι θα γίνει ενημέρωση, επικαιροποίηση το 2014 να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τις σχετικές εγγύησεις για τον τομέα του ηλεκτρισμού και έχουμε διάφορους τομείς εδώ στον τομέα των μεταφορών οπότε να έχουμε μια εργαλειοθήκη πλήρη με όλα αυτά τα μέσα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε σχέση με το Connecting Europe Facility. Δεν λέμε τώρα την τεχνική αρρωγή, πάντως πρόκειται για πολύ βασικό χαρακτηριστικό και στοιχείο αυτής της εργαλειοθήκης. Πάμε τώρα παρακάτω. Μιλήσαμε για την κατανομή των ε, στοιχείων του προπολογισμού και τώρα συνάδελφος θα συνεχίσει. Τζόρτζιου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας αυτή. Θα μπορέσω κατά αυτόν τον τρόπο να σα ενημερώσω για την πρωτοβουλία των ομολογιακών δανείων για τη χρηματοδότηση έργων. Ξέρω ότι το ζήτημα αυτό ορισμένοι το έχετε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Πάντω, πολύ σύντομα να σα πω ότι πρόκειται για ένα κοινό πρόγραμμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει χρηματοδοτικά κάποια ομολογιακά δάνεια, κάποια έργα, προκειμένου να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε τα ομόλογα αυτά στις ε, αγορές, στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις παγκόσμιες αγορές και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε άμεση χρηματοδότηση από την αγορά, από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, από ασφαλιστικούς για παράδειγμα οργανισμούς, προκειμένου να χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα έργα στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Την τελευταία φορά που σα δώσαμε κάποιε πληροφορίε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από έξι μήνε περίπου, σα είχα πει ότι ήμασταν τότε σχεδόν έτοιμοι να υπογράψουμε το δεύτερο πρόγραμμα, αν θέλετε, το δεύτερο τέτοιο έργο το οποίο θα εμφανίζεται στην κοινή αυτή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όσον αφορά δηλαδή συγκεκριμένα έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο Βέλγιο. Σας είχα πει τότε ότι θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας παρουσιάσω ένα ακόμα έργο. Ένα έργο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ένα ακόμα έργο το οποίο αφορά τις ειδικές συναλλαγές. Τα έχουμε πετύχει αυτά και τα δύο και θα στα παρουσιάσω αυτή τη στιγμή. Όσοι τώρα ενδιαφέρονται να καταλάβουν λίγο περισσότερο πώς λειτουργούν τα μέσα αυτά από τεχνικής πλευράς, μπορώ κατηνδίαν επίσης να σας δω και επίσης έχω και ένα σύντομο έγγραφο μαζί μου το οποίο περιγράφει ακριβώς το πώς διαρθρώνται τα έργα αυτά και πώς λειτουργούν σε τεχνικό επίπεδο. Ας περάσουμε τώρα στα project αυτά καθ' αυτά, στα έργα τα οποία έχουμε στην κοινή αυτή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η πρώτη, αν θέλετε, συναλλαγή είναι το Greater Gatboard Offshore Transmission Project, Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο στον Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει να κάνει με υπεράκτιες πλατφόρμες ενέργειας, ένα έργο το οποίο εμφανίζεται λοιπόν στην κοινή αυτή συμφωνία που έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων και όπου χρησιμοποιήθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να βαθμολογήσουμε το έργο αυτό στις παγκόσμιες αγορές με το βαθμό α πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε με πολύ χαμηλά επιτόκια το έργο αυτό και από ό,τι φάνηκε ε, εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τρεις φορές ε, μεγαλύτερο από ό,τι περιμέναμε από διάφορους επενδυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ πέρα είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή συναλλαγή. Το δεύτερο έργο, η δεύτερη συναλλαγή, την οποία ήθελα να σας παρουσιάσω την προηγούμενη φορά που είχα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αυτή που έχει να κάνει με τον αυτοκινητόδρομο Α11 στο Βέλγιο, ο πρώτος, αν θέλετε, οικολογικός αυτοκινητόδρομος, έργο το οποίο υπεγράφει το Μάρτιο του 2014. Στην περίπτωση αυτή είχαμε 150 εκατομμύρια μέσω ομολογιακών δανείων που υποστηρίζουν ένα συνολικό ποσό 580 εκατομμυρίων. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το τμήμα, το ποσοστό εκείνο το οποίο έχουμε μέσω ομολογιακών δανείων. Και έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στο έργο αυτό. Καταφέρνουμε να αντλήσουμε περισσότερα κεφάλαια από επενδυτές και μάλιστα τα κεφάλαια αυτά είναι μακροχρόνια, κάτι το οποίο σπάνια συμβαίνει στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου η χρηματοδότηση είναι συνήθως βράχη πρόθεσμη. Το καλοκαίρι του 2014 υπογράψαμε το πρώτο έργο το οποίο έχει να κάνει με τις τηλεπικοινωνίες Αξιώνε Infrastructure Γαλλίας. Υπεγράφει λοιπόν το έργο αυτό και είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα 20 εκατομμύρια τα οποία έχουμε από τα κοινοτικά ταμεία όσον αφορά τα έργα τηλεπικοινωνιών. Ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που είχαμε για τον κλάδο αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε τα πρώτα μέσα Χρηματοδότηση των έργων αυτών από τις παγκόσμιες αγορές είχαμε ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα. Καταφέραμε να αντλήσουμε 38 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων, φτάνοντας ένα συνολικό ποσό 190 εκατομμυρίων ευρώ για ενδεκαετή περίοδο, έχοντας επίσης πάρα πολύ καλές ευνοϊκές τιμές και ευνοϊκά επιτόκια για ένα έργο στο οποίο ουσιαστικά ο ιδιωτικός τομέα αναλαμβάνει ένα κάποιο βαθμό κινδύνου. αν θέλετε, η τιμή για το έργο αυτό ήταν ιδιαίτερα πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τη τιμή που θα είχε το έργο αυτό αν είχε απλώς χρηματοδοτηθεί απλώς μέσω μιας τράπεζας. Το πιο πρόσφατο έργο το οποίο υπεγράφει τον Αύγουστο του 2014 είναι η δημιουργία του αυτοκινητοδρόμου Α7 στη Γερμανία. Πάλι εδώ πέρα προβλέπεται μια συμφωνία χρηματοδότηση του έργου αυτού με ένα σημαντικό το ποσό μόχλευση 68 εκατομμύρια ευρώ μέσω εμαλογιακών δανείων που υποστηρίζουν ένα γενικότερο ομόλογο 725 εκατομμυρίων ευρώ. Πάλι εδώ πέρα οι συνθήκε οι τιμολογιακέ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και θεωρούμε ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται κατά τρόπο πολύ πιο ανταγωνιστικό αν να συγκρίνουμε τη χρηματοδότησή του με τις πιο παραδοσιακές μορφές ε, χρηματοδότησης. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα όσον αφορά το σύστημα πληροφορική που χρησιμοποιούμε, είναι λίγο παροχημένο. Τώρα όσον αφορά το τέλο του έτου, στα τέλη του 2014, Θεωρούμε ότι τρία ακόμα έργα θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του 2014 στην Ιταλία και στην Ιρλανδία συγκεκριμένα, δύο νέες χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία ομολογιακών έργων. Θα έχουμε επίσης ένα ακόμα έργο και στη Γαλλία στον τομέα των μεταφορών. Κατά τα λοιπά, είπαμε ότι αυτή η πιλωτική φάση θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2016, οπότε τα έργα θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την, την ΕΤΕ μέχρι τα τέλη των εστώτος έτους, οπότε θα έχουμε και να ολοκληρώσουμε το τέλος του 2016 και προς το παρόν βλέπετε ότι έχουμε 216 εκατομμύρια από τέτοιου κεφάλαια ε, κεφάλαιο το οποίο πρόκειται να βοηθήσει αυτά τα προγράμματα και θα μας οδηγήσει σε κάποια ομόχλευση μέχρι το ύψος του 1,3 ε, εκατομμύριων από αυτά τα 7 δις ε, συνόλου των δανείων και ομολόγων. Οπότε βλέπετε πώς θα μπορέσουμε με τα ομόλογα αυτά να υποστηρίξουμε αυτά τα προγράμματα και αυτές είναι οι άμεσες προοπτικές. εν κατακλείδη. Αναμφίβολα ενδιαφέρεται πάρα πολύ η αγορά για αυτού του είδους την πρωτοβουλία και θεωρείται ότι έτσι θα χρηματοδοτηθεί η υποδομή στην Ευρώπη. Τα έργα υποδομής και έτσι θα έχουμε μια καινούργια πηγή χρηματοδότησης στα έργα υποδομής στην Ευρώπη. Οπότε θα έχουμε τώρα περισσότερες επιλογές πέραν της παραδοσιακής ε, τραπεζικής πηγής θα έχουμε τα τα ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και έτσι θα μπορέσουν όλοι αυτοί άμεσα να χρηματοδοτήσουν. Η ανταπόκριση επομένως ήταν ε, άμεση, ήταν ισχυρή πέραν της ε, προσθέμενης αξίας που έχουμε από αυτά τα ομολογιακά ε, δάνεια και για να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε Λέμε ότι υπάρχει ισχυρό έντονο ενδιαφέρον για αυτή την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε ότι ο στόχος των 5 7 προγραμμάτων για αυτή την πυρογική φάση θα την πετύχουμε και θα υπάρξει αντίκτυπος πάρα πολύ σημαντικός η ανταπόκριση από τους εταίρους μας, από τους επενδυτές είναι ενδιαφέρον. Ακόμα βέβαια θα πρέπει να ενδιαφερθεί περισσότερο το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει το δημόσιο να αλλάξει κάπως τους διαγωνισμούς και να είναι αυτή πιο φιλική ούτως υπήν προς αυτά τα ομολογιακά δάνεια. Πάντως βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά και σε έξι μήνες πρόκειται να σας ενημερώσουμε και πάλι για το πώς θα συνεχιστεί η πορεία αυτής της πρωτοβουλίας. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σαφέστατη αυτή παρουσίαση που πραγματικά αποδεικνύει την επίπτωση μόχλευσης που έχουν τα ομολογιακά αυτά δάνεια. Ως προς τον προπολογισμό όμως ποιος θα είναι ο αντίκτυπος. Ξέρουμε ότι πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κάποια εγγύηση, έτσι δεν είναι. Τα πρώτα χρόνια νομίζω τα πράγματα εξελίσσονται πολύ θετικά. Αν όμως, Φερρυπίν, κάποια στιγμή ένας επενδυτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες του, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει όπως είχε πει στην αρχή, ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μας το αυτό να απαντήσω στην ερώτηση αυτή άμεσα. Τα 230 εκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιούνται από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο στάδιο είναι μια συμβολή κεφαλαιακή που γίνεται από τον κοινοτικό προπολογισμό προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να καταφέρουμε να, καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες, τις πρώτες χρηματοδοτικές ανάγκες και να δοθεί μια πρώτη, αν θέλετε, εγγύηση για, την, για το πρώτο τμήμα χρηματοδότησης των έργων. Κατά αυτόν τον τρόπο, με τα χρήματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να προκαταβάλει κάποια ποσά και μπορεί να εκδώσει αυτά τα ομολογιακά δάνεια. Και στη συνέχεια, η το ομολογιακό δάνειο εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν προκύψει λοιπόν κάποιο πρόβλημα όπως είπατε, τότε το χρέος αυτό το οποίο καλύπτεται από μία εγγύηση ή από μία μερική εγγύηση, τότε εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να καλύψει το κενό που ενδεχομένω προκύψει από του δικού τη του πόρου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να κάνει όμω κάτι τέτοιο, γιατί αν δούμε το σύνολο των έργων, το σύνολο του χαρτοφυλακίου δηλαδή, οποιαδήποτε απώλεια μπορούμε να έχουμε από τα πρώτα 230 εκατομμύρια ευρώ, έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επηρεάζεται όμω ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιαδήποτε μελλοντική απώλεια. Το μόνο το οποίο ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πρώτη φάση είναι αυτά τα 230 εκατομμύρια ευρώ. Οποιαδήποτε απώλεια ή χρέωση οφειλεί προκύψει στη συνέχεια, αυτό αποτελεί πλέον ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ακριβώ επειδή λειτουργούμε σε συνθήκες, πραγματικές συνθήκες της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδη λειτουργουμε σε συνθηκες πραγματικες συνθηκες μπορεί και να αποζημιωθεί για τον κίνδυνο το οποίο αναλαμβάνει. Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί κανένα ευρώ από τα 230 εκατομμύρια ευρώ και θα κερδίσει μάλιστα και σε απόδοση, η, σε απόσβεση δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χειρότερη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν τα ποσά αυτά, 230 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, και πάλι όμως την ευθύνη θα αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξ ολοκλήρου. Πάντως στο έγγραφο το, αυτό το οποίο σας παρουσίασα παρουσιάζουμε πραγματικά όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας για πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώσουμε στη μία παρά 20. Ποιο θέλει το λόγο παρακαλώ. Ουδής. Eh Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τη συνεδρίασή μα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά ήσασταν σαφέστατοι στις παρουσιάσεις που κάνατε. Βλέπουμε πραγματικά ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα υψηλότατο επίπεδο μόχλευσης, ότι απορρέουν πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες μέσω των ομολογιακών αυτών δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων και θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε εν μέρη τα 307 δισεκατομμύρια στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Γιούνκερ στο λόγο τον οποίο εκφώνησε λίγα λεπτά μετά την επίσημη εκλογή του θα έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε εκ νέου το ζήτημα αυτό, το πιο σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ποιο θα είναι ο δημοσιονομικό αντίκτυπο των ομολογιακών αυτών δανείων στον κοινοτικό προπολογισμό. Κύριε Ντεπρέ, όπως καταλάβατε, θα πάρετε το λόγο για, τα, για τους διορθωτικούς προπολογισμούς του 2014 στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Κύριε Ντεπρέ, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα έχω απλώς, κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι πολύ καλά ότι είχα ήδη παρουσιάσει τα όσα έχουν να κάνουν με τους διαρθετικούς προπολογισμούς υπαριθμών 2, 3 και 4 κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Ιούλιο. Νομίζω ότι ήμουν απόλυτα σαφής τότε, είχα εξηγήσει τα πάντα και σας είχα πει ποια θα ήταν η πολιτική στρατηγική την οποία είχαμε τότε εγκρίνει. Είμαι λοιπόν στην διάθεση της Ευρωπαϊκής, ε, μάλλον συγγνώμη, είμαι στη διάθεση της Επιτροπής μας για να απαντήσω σε επιπλέον ερωτήσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι εντελώς περιττό αυτή τη στιγμή να επαναλάβω τα όσα πολύ σαφέστατα σας είχα πει στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά στη διάθεσή μας, λέει ο Πρόεδρος. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενδεχομένως να προκύψουν και κάποια προβλήματα. Ορισμένες αρχές μπορούν να θεωρούν ότι το πλεόνασμα του 2013 θα πρέπει ουσιαστικά να επιστραφεί στα κράτη-μέλη. Εσείς πάντως μας είπατε ότι το πλεόνασμα του 2013 είναι καθαρά θεωρητικό. Για το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε πάρα πολύ το ποσό των μη εξοφλημένων πληρωμών. Άρα δεν μιλάμε πραγματικά για πλεόνασμα, έτσι δεν είναι αν ήταν πραγματικά προσεκτική και επιμελής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είχε χρησιμοποιήσει το πλεόνασμα αυτό προκειμένου να εξοφλήσει τις πληρωμές που δεν είχαν ακόμα καταβληθεί. Ο κύριος Δεπρές, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Πρόεδρε. Τα νομικά κείμενα όμω υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο να υποβάλει ένα συγκεκριμένο έγγραφο όσον αφορά τα πλεονάσματα τα οποία προκύπτουν από το προηγούμενο έτο. Πρόεδρο, ναι, θα ήθελα απλώ όμω να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εκμεταλλευτούν την περίπτωση αυτή τα κράτη-μέλη προκειμένου να ζητήσουν επιστροφή των κονδυλίων αυτών στου εθνικού προπολογισμού, να μην χρησιμοποιήσουν κατά αυτόν τον τρόπο το πλεόνασμα 2013. Μα συμφωνώ μαζί σα, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Δεπρέ, γι' αυτό ακριβώ υιοθετήσαμε την ακόλουθη στρατηγική. Να ομαδοποιήσουμε τις προτάσεις διορθωτικών προπολογισμών 2, 3 και 4 και να καταλήξουμε σε ένα συνολικό ποσό το οποίο να μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε σε κοινοτικό επίπεδο. Έχετε επίσημη συμφωνία γι' αυτό όμως, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Υπάρχει κάθε νόημα το πλεόνασμα ενός έτους να μπορούσε να λειτουργήσει ως μια συνταγή και να περάσει ως έσοδα και να περάσουν αμέσως στο επόμενο έτος και να μην είναι πίστοση για κάθε κράτος μέλος. Και ερωτώ, αν αυτό το πνεύμα έτσι με αυτόν τον τρόπο αντανακλάται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον κανονισμό του. Και έτσι σε σχέση με, τον, με το περιθώριο να μπορούσε να, να λειτουργήσει δηλαδή μετάβαση από το ένα έτος προς το άλλο μέχρι συγκεκριμένα ποσά, μέχρι συγκεκριμένο ύψος ποσών. Η ερώτησή μου λοιπόν διατυπώνεται ως εξής. Υπάρχει κάποιος τρόπος ή μπορεί έτσι να καθιερωθεί ότι τα, πλεονάσματα θα μπορούν να είναι έσοδα του επόμενου έτους. Ευχαριστώ. Το μικροφόνο Πρόεδρος. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι μία παρά 20 και πρέπει υποχρεωτικά να σταματήσουμε. Θα απαντήσουμε στη συνέχεια στην ερώτηση σε αυτή. Φοβάμαι ότι απάντησαν αρνητική. Λοιπόν, συνεχίζετε πάλι στην ιδρύσή μας στις 3 το μεσημέρι.